Ξεκινάμε. Benvenuti a tutti. Καλώς ορίσατε όλοι. Benvenuti a tutti. Καλώς ορίσατε όλοι. Ξεκινάμε, όλοι ξεκινάμε τη συνεδρία της Επιτροπής. Ολοκληρώσαμε τη συνεδρία των συντονιστών. Θα ενημερωθείτε από τους συντονιστές σας για τα νέα. Περνάμε στο σημείο 2, υιοθέτηση της ημερήσιας διάταξης. Ο εισηγητής μα ε, για τα μέτρα που αφορούν συγκεκριμένα το τομέα τη γεωργίας της άκρως απομακρυσμένε περιοχές ε, δεν θα μπορέσει, ο κύριο Αντρόβερ, Αντρόβερ δεν θα μπορέσει να βρίσκεται εδώ αύριο το πρωί, συνεπώ. θα χρειαστεί να αναβάλουμε το σημείο 7 τη υπηρεσία διάταξη, Αλλά ο αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριο Γιώργο Παπαστάμκο, έκανε το ίδιο αίτημα. Έτσι λοιπόν και το σημείο 8, καθορισμό ειδικών μέτρων για τη Γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου, θα αναβληθεί. Τα σημεία λοιπόν 7 και 8 της ημερήσιας διάταξης θα αναβληθούν για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 26-27 Νοεμβρίου. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη με αυτήν την τροποποίηση. Σας ενημερώνω ότι σήμερα μας λείπουν κάποιες γλώσσες. Πιο συγκεκριμένα λείπουν τα φιλανδικά, τα λιθουανικά και τα σλοβένικα. Ζητώ λοιπόν συγγνώμη για αυτό το πρόβλημα. Σας ενημερώνω ε, ε, επιπλέον ότι η σημερινή συνεδρίαση μεταδίδεται με web streaming στις 13 επίσης Νοεμβρίου. Δώστε λίγο προσοχή. Στις 3 ώρα το απόγευμα, από τις 3 ώρα το απόγευμα μέχρι τις 6 η Επιτροπή Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Επιτροπή ΙΜΚΟ και τη δική μας Επιτροπή θα διοργανώσει μια ακρόαση με τον επίτροπο που όρισε η Μαλτέζικη κυβέρνηση για την υγεία των καταναλωτών, τον κύριο Μπόργ, Αντώνιο Μπόργ. Οι συντονιστές μας θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήσεις σε σχέση με τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας. Όπως αποφασίσαμε μεταξύ συντονιστών, θα υποβάλουμε πέντε ερωτήσεις, μία από κάθε ομάδα. Ήθελα επιπλέον να σας ενημέρωσω, όπως αποφασίσαμε μεταξύ συντονιστών, ότι αποφασίσαμε να αναστείλουμε την ψηφοφορία για τις εκθέσεις, για τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής για τις 23-24 Ιανουαρίου του 2013. Όπως γνωρίζετε υπάρχει ανάγκη να μεταφραστούν όλες οι συμβαστικές τροπολογίες σε όλες τις γλώσσες και αυτό οδηγεί σε αναστολή, αναβολή για τις 23-24 Ιανουαρίου που είναι η τελική ημερομηνία. Αυτό σημαίνει ότι οι δικοί μας εισηγητές θα πρέπει να υποβάλουν τα κείμενα των συμβιβαστικών τροπολογιών για μετάφραση ενδεχομένως έως τις 15 Δεκεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση πριν από τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές ώστε να έχουμε μεταφρασμένα τα κείμενα στη... και για να τα συζητήσουμε 23 και 24 Ιανουαρίου. Ελπίζουμε ότι 23-24 Ιανουαρίου θα μπορέσουμε να προβούμε και σε τελική ψηφοφορία εφόσον έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση για τις δημοσιονομικές προοπτικές. Σημείο 4. Έγκριση των πρακτικών ε, των ε, συνεδριάσεων της 3 Σεπτεμβρίου και της 17 18 Σεπτεμβρίου. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, τα πρακτικά λοιπόν εδώ θα, θεωρηθούν ότι έχει, θα θεωρηθεί ότι έχουν εγκριθεί. Περνάμε τώρα στο σημείο 5, Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Εισηγητή σύντακτη γνωμοδότησης Λουίς Παύλο Αλβές που βρίσκεται εδώ και τον οποίο χαιρετίζω. Ξεκινάμε λοιπόν τη συζήτηση εδώ με την ψηφοφορία για αυτό την έκθεση. Είχαμε ορίσει για σήμερα την ψηφοφορία ώστε η αρμόδια επιτροπή ε, επί της ουσίας που ήταν η Επιτροπή ΕΜΠΛΕ να μπορέσει να υιοθετήσει την έκθεση της αύριο λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις μας. Πριν δώσω το λόγο στον συντάκτη κύριο Άλβες ήθελα να σας ε, να επιστήσω την προσοχή σας ε, στην λίστα ψηφοφορίας. Έχουμε τρεις τύπους τροπολογιών. Πρώτον, έχουμε τις τροπολογίες που αποσκοπούν στον αποκλεισμό των γεωργών από την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Δεύτερον, υπάρχουν τροπολογίες που διατηρούν την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους γεωργούς και τροποποιούν συνεπώς τις διατάξεις όσον αφορά τους γεωργούς και τρίτον, τρίτο είδος ε, τροπολογιών. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που δεν έχουν σχέσεις με τις συγκεκριμένες διατάξεις που αφορούν τους γεωργούς και συνεπώς είναι συμβατές με τους άλλους δύο τύπους τροπολογιών. Επειδή οι πρώτοι δύο τύποι δεν είναι συμβατοί μεταξύ τους, θα έχουμε δύο μαζικές ψηφοφορίες στην αρχή. Το αποτέλεσμα αυτών των δύο πρώτων ψηφοφοριών θα ορίσει κατά πόσο θα ζητήσουμε από την Επιτροπή ΕΜΠΛ να αποκλείσει τους γεωργούς από αυτόν τον κανονισμό του ή όχι. Νομίζω ότι σας παρουσίασα αυτή τη στιγμή ε, συνοπτικά τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε. Τώρα θα ήθελα να δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο εισηγητή. Δεδομένου ότι μας ανακοινώθηκε και μια προφορική τροπολογία, θα ακούσουμε και την προφορική τροπολογία στη συνέχεια. Λουίς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε ενώπιον μας μία γνωμοδότηση που θα επιδώσουμε στην Επιτροπή Απασχόλησης με θέμα το κατά πόσο θα συμπεριληφθούν ε, ή όχι οι γεωργοί στο Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Αυτό όμως δεν είναι το μόνο θέμα. Γιατί από την ε, ψηφοφορία μας δεν θα προκύψει νομοποίηση για να συμπεριλάβουμε τελικά τους γεωργούς σε αυτό το ταμείο. Και αυτό βάρινε πολύ στον τρόπο που κατήρτισα την γνωμοδότησή μου. Μια και η Επιτροπή μας δεν έχει την ικανότητα να συμμετέχει στη συζήτηση για να προσπίσει τα δικαιώματα των γεωργών, τελικά συνέταξα την γνωμοδότησή μου υπερασπίζοντας τη θέση ότι ελήψη καλού εργαλείου που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μια και το το Ταμείο αυτό με τον κανονισμό δεν μας επιτρέπει να προσπίσουμε δεόντως τα συμφέροντα των Γεωργών. Τελικά, ε, το ότι δεν περιλαμβάνονται στον κανονισμό ε, ίσως είναι καλύτερο, γιατί αν συμπεριληφθούν στον κανονισμό θα θεωρηθεί από μερικού ότι ε, δικαιούνται ή τη χάνουν μιας προστασίας που σε τελική ανάλυση δεν θα απολαύσουν. Η γνωμοδότησή μου αυτή τη θέση ουσιαστικά υποστηρίζει. Ότι ο κανονισμός δεν είναι προσαρμοσμένος στις καταστάσεις και προτιμούμε να διεκδικήσουμε αυτά τα κονδύλια σε ένα καλύτερο πλαίσιο της κοινή γεωργικής πολιτικής για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν καλύτερα για τους γεωργούς. Ευχαριστώ. Ωραία. Ας προχωρήσουμε. Έχετε όλοι τις κάρτες ψηφοφορίας σας. Ξεκινάμε την ψηφοφορία. Μαρία ζητάει το λόγο. Εγώ δεν έχω την κάρτα ψηφοφορίας μου επειδή είναι Δευτέρα. Παρακαλώ να με υπολογίσετε. Ευχαριστώ. Ωραία λοιπόν και ο Λούις ε, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Πρώτα απ' όλα ψηφίζουμε μαζικά την πρώτη ομάδα λοιπόν τροπολογιών. Τροπολογία 12 Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Πρέπει να μετρήσουμε ποιος είναι υπέρ. Ψήφισαν όλοι. Το μηχάνημα δεν λειτουργεί εκεί. Θα πρέπει να υπολογίσουμε και τον Αντιπρόεδρο. Εδώ λειτουργεί τώρα, ζητώ συγγνώμη, δεδομένου ότι είναι σημαντική αυτή η ψηφοφορία. Α επαναλάβουμε. Πάτρε, ξεκινάμε από την αρχή. Επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίστε όλοι. Και μετά όσοι δεν έχουν κάρτα, ας μας το επισημάνουν. Πέρας της ψηφοφορίας. Πόσοι δεν έχουν καρτέλα. Εσύ ψήφισες με την κάρτα. Και απήχε και... Νο, όχι. Τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ε, είναι ότι απορρίπτεται. Όχι. να ελέγξουμε ε, Αυτά το 18-17 είναι ηλεκτρονική ψηφοφορία αλλά λαμβάνουμε υπόψη και τα τρία μέλη που δεν έχουν τις κάρτες τους. και 18 18-18 αυτό σημαίνει απόρριψη. Ναι, ήταν 18-17 και 2 κατά. Λοιπόν, 19-19 σημαίνει ότι απορρίπτεται. Ας προχωρήσουμε λοιπόν. Περνάμε στην τροπολογία τώρα αριθμός 9. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την τροπολογία 9. Είμαστε βέβαιοι ότι δεν υπάρχουν και άλλα μέλη του ΕΛΚΑ. Είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει ένας παραπάνω του ΕΛΚ. Είκοσι με 19 τελικά, λέει ο Πρόεδρος, ήταν, ξεκινά η ψηφοφορία για την τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 9. Παρακαλώ ψηφίστε για την τροπολογία 9. Κυρία Μαγκίνες, αυτή τη φορά θα ψηφίσω με την κάρτα μου για να το διευκρινίσω για τους συναδέλφους. Ωραία η κυρία Μαγκίνες έχει την κάρτα ψηφοφορίας. Ψηφίστε όλοι για τροπολογία 9. Κλείνει η ψηφοφορία. 18. 18. Ποιος δεν έχει την κάρτα ψηφοφορίας. Καλινόσκι και και Καπούλας είναι υπέρ, Καλινόσκι είναι κατά 19-19, Σεγκρέσκι είναι, Σιλβέστρη είναι κατά. Συνεπώ, απορρίπτεται. Έχουμε τώρα την προφορική τροπολογία. Ποιος θα την παρουσιάσει. Νικολέσκου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το κείμενο της προφορικής τροπολογίας ε, σας το έχουμε μοιράσει. Δεν πρόκειται να το διαβάσω, απλώς θα ήθελα να διευκρινίσω ότι οι δύο προφορικές τροπολογίες έχουν τον ίδιο στόχο. Δηλαδή, την διαγραφή της φράσης με βάση τις εμπορικές συμφωνίες που αφορούν την γεωργία. προτιμούμε να μιλούμε για τους δικαιούχους ε, της, ε, του ταμείου αυτού. Αυτό είναι ο στόχος των δύο τροπολογιών. Ευχαριστούμε πολύ, αξιότιμο κύριε Νικουλέσκου. Πρέπει να ρωτήσω, αντιτίθεται κανείς, έχει αντίρρηση με αυτές τις προφορικές τροπολογίες. Με αυτή την προφορική τροπολογία κανείς δεν είναι αντίθετος. Ναι. Υπάρχουν αντίθετοι ο εισηγητής. Όχι. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν αντιρρήσει. Σύμφωνα με τον κανονισμό, αν υπάρχουν αντιρρήσει, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε για την προφορική τροπολογία. Προχωράμε τώρα με τι τροπολογίε. Με την τροπολογία 49 Μαγκίνε άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 49. Άρχεται η ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 48 της κυρίας Λούλινγκ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέρμα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Την τροπολογία νούμερο 10 του κυρίου Συγητή. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 54 στην επόμενη σελίδα. Άρχεται η ψηφοφορία για την 54. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία. Στη συνέχεια ψηφίζουμε την τροπολογία. 56. Μαγκίνες. Άρχεται η ψηφοφορία για την 56. Ψηφίσατε όλοι. Ναι. Πέρας ψηφοφορίας. Αγκρίνεται. Περνάμε στην ψηφοφορία για την τροπολογία 59. Νικουλέσκο, Άρχεται η ψηφοφορία. 59. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 60. Άρχεται η ψηφοφορία για την 60. Ψηφίστε για την τροπολογία 60. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 62. Λαβία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 63, Πατράων Εβές. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 64. Σιλβέστρης. Άρχεται η ψηφοφορία. 64 τροπολογία. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Περνάμε στην 67 Πατράων Εβές. Άρχεται η ψηφοφορία. 6 67 67. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Περνάμε στην ψηφοφορία τώρα για την τροπολογία 68 Μαγκίνες. Άρχεται η ψηφοφορία για την 68 πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η 68. Περνάμε στη συνέχεια στην 69 Νικουλέσκου. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 71 Πατράων Εβές. Άρχεται η ψηφοφορία. 71 τροπολογία. Ψηφίσατε όλοι για την 71. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην 22. Άρχεται η ψηφοφορία για την 22. Ψήφισατε όλοι για την 22. Εγκρίνεται. Με μεγάλη διαφορά. 23 ψηφίζουμε τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 72. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την 72. 72. Προσοχή. Ψηφίσατε όλοι για την 72. Πέρας ψηφοφορία, Απορρίπτεται. Περνάμε στην 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα για την 74. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 74. Ψηφίστε για την 74. Ψήφισαν άπαντες. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 75. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε άπαντες. Απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 29 Λούλινγκ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Και απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 3. Πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 3. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 3. Για το εκτιμώντας 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 3. Αιτιολογική σκέψη 5. Τροπολογία 3 του εισηγητή. Ψηφίσατε άπαντες. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Περνάμε μετά στην 37 Νικουλέσκου. Άρχεται η ψηφοφορία για την 37 του κυρίου Νικουλέσκου. Ψήφισαν όλοι. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα Πρέπει να ψηφίσουμε τώρα την 39. Ζητώ συγγνώμη, αλλά είναι περίπλοκα τα πράγματα σήμερα. 39. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την τροπολογία 39 πατράουν Εβέ. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Περνάμε τώρα. «43». Τροπολογία 43. Πατράων Πατράω Νεβές. Άρχεται η ψηφοφορία για την 43. Κλείνει η ψηφοφορία για τη 43 και απορρίπτεται. Περνάμε στη 44. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 44. Πέρας ψηφοφορίας για τη 44 και απορρίπτεται. Και περνάμε στη 45. Το ίδιο. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 45. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην τελευταία τροπολογία νούμερο 47. Ψηφίζουμε τη 47. Τελευταία τροπολογία. Ψηφίσατε άπαντες. Απορρίπτεται. Ψηφοφορία για το σύνολο της γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία για το σύνολο της γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Προσοχή. Υπέρ. Εδώ είναι ενδιαφέρουσα πολύ η τελική ψηφοφορία για την γνωμοδότηση όπως τροποποιήθηκε. Είναι εδώ όλοι, έχουμε όλες τις κάρτες ψηφοφορίας, έχετε ψηφίσει άπαντες. Απορρίπτεται. Όχι, όχι, τι... 16 αποχές, απορρίπτεται. Τελικό αποτέλεσμα είναι ότι η Επιτροπή μας δεν έχει άποψη για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση. Κύριε Άγνιου, ζητήσατε το λόγο. Απλά για προς όφελος των όσων ξέχασαν ε, ή έχασαν τις ε, κάρτες ψηφοφορίας τους δεν μπορείτε να λάβετε νέα από το γραφείο κάτω από την αίθουσα της Ολομέλειας. Όλα αυτά έχουν κλείσει. Χρειάστηκα 25 λεπτά για να το μάθω σήμερα το απόγευμα για να πάρετε μια άλλη κάρτα ψηφοφορία πρέπει να πάτε στο τέλο των pigeonholes των βουλευτών. Εκεί υπάρχει ένα γραφείο και εκεί μπορείτε να λάβετε άλλη μια νέα κάρτα ψηφοφορία. Okay, Ωραία, ευχαριστούμε τον κύριο Άγνιο. Η ψηφοφορία όμως ήταν σαφής. Η Επιτροπή μας δεν έχει άποψη για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 6. Παρουσίαση της μελέτης με θέματα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσίαση μελέτης μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενθάρρυνση και την υποστήριξη των εισερχομένων. Θα ήθελα να δώσω το λόγο και να καλωσορίσω τον κύριο Χέσους Κονσάλες ε, Ρεχιντόρ από το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο, τον Εξάρτητο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης που θα μας παρουσιάσει μια μελέτη για τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενθάρρυνση και την υποστήριξη των νέων εισερχομένων. Όποιος θέλει να καταλήψει την αίθουσα μπορεί, αλλά παρακαλώ ήσυχα. Παρακαλώ σταματήστε τη συζήτηση εντό τη αίθουσα. Δίνω το λόγο στον κύριο Χεσού Ρεχιδόρ από το, αυτόνομο, από το Ανεξάρτητο Πανεπιστήμιο τη Μαδρίτη να μα παρουσιάσει αυτή τη μελέτη που μα ενδιαφέρει για τι ενιαίε ενισχύσει και τα ζητήματα που εξετάζουν οι σκιώδει συζητητέ όσον αφορά αυτό το φάκελο. Δίνω λοιπόν το λόγο ζητώντας συγγνώμη για αυτό το σαματά Ζητώ συγγνώμη κύριε Γκοντζάλε, αλλά ήταν λίγο περίπλοκη η ψηφοφορία. Έχετε το λόγο για να μα παρουσιάσετε την έκθεση. minutes. 15 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που μου δίνεται ευκαιρία να παρουσιάσω τα βασικά πορίσματα μιας έκθεσης που πολύ πρόσφατα ολοκληρώθηκε, μιας μελέτης για τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν προκειμένου να δοθούν κίνητρα και ενάψματα για την ε, ανάληψη γεωργικών δραστηριοτήτων από νέου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ε, διαπιστώνετε κι εσείς, είναι ένα θέμα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής για πολλούς και διάφορους λόγους, τους οποίους ε, θα σας αναλύσω στη συνέχεια. Το θέμα των εισορχομένων στη Γεωργία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια και η κοινή γεωργική πολιτική περνάει από μια νέα διαδικασία μεταρρύθμισης. Θα ήθελα λοιπόν να σας σχολιάσω πρώτα απ' όλα το σημείο κίνησης αυτού του προβλήματος, ποια ήταν η αφετηρία του και να σας δώσω εν συντομία κάποια στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση που σας προανέφερα. Στην έκθεση μάλιστα αυτή περιλαμβάνονται πολλές στατιστικές πληροφορίες και στοιχεία αναχώρα. Και στο σκαρίφημα που σας μοίρασα ε, δεν ε, υπάρχουν τα παραρτήματα, αλλά στην οριστική εκδοχή της έκθεσης θα συμπεριληφθούν και τα παραρτήματα με αναλυτικά στοιχεία για όλες τις χώρες. Τα παραρτήματα αριθμών 20 και σελίδε, θα βρείτε εκεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Θα ήθελα όμω συνοπτικά να τονίσω τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία που δείχνουν τη σοβαρότητα του προβλήματο που αντιμετωπίζουμε. Θα ήθελα να πω καταρχήν ότι το θέμα της έλλειψης ή της σπάνιας των νέων γεωργών ε, παρατηρείται σε ένα πλαίσιο που εδώ και καιρό χαρακτηρίζεται από σταδιακή μείωση του αριθμού και των γεωρικών εκμεταλλεύσεων και των γεωργών. Πρόκειται για μια διαδικασία που τα τελευταία χρόνια επιταχύνθηκε. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον αριθμό των γεωργών. Μειώνεται σταδιακά λοιπόν ο αριθμό των γεωργών. Και για να διαμορφώσετε μια συγκεκριμένη άποψη για τη σοβαρότητα του προβλήματο, θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι μόλι το 6% των ε, γεωργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι αυτή τη στιγμή κάτω των 35 ετών. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Μόλις το 6% των Ευρωπαίων Γεωργών ε, είναι κάτω των 35. Το 5% στην, ε, στις 15 χώρες και 7% στις 12 χώρες της, ε, της τελευταίας διεύρυνσης. Η άλλη όψη του νομίσματος αφορά την κατάσταση των πιο ηλικιωμένων γεωργών που είναι 55 ετών και άνω, που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 55% του συνόλου των γεωργών. Έχουμε μια, ε, ένα μικρό αριθμό νέων γεωργών και ένα γυράσκοντα γεωργικό πληθυσμό. Πάνω από το 55% των Ευρωπαίων γεωργών, επαναλαμβάνω, είναι άνω των 55 ετών. Και αυτό είναι πολύ πιο σοβαρό και πιο οξύ το πρόβλημα στις 15 παλιότερες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης από ό,τι 12 ε, της νέας διεύρυνσης, όπου το, πρόγραμμα είναι, το πρόβλημα είναι λιγότερο οξύ. Θα ήθελα τώρα να χρησιμοποιήσω ένα δίκτυ που αφορά το ποσοστό της αντικατάστασης των γεωργών. Των κατόχων, δηλαδή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, των holders. Διαπιστώνουμε αυτό το ποσοστό αντικατάστασης που είναι κατά κάποιο τρόπο η εγγύηση ότι θα υπάρξει κάποιο γεωργό που θα συνεχίσει τη γεωργική δραστηριότητα, βλέπουμε ότι το ποσοστό αυτό τη αντικατάσταση ανέρχεται μόνο στο 15% στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 χωρών μέλων, των πρώτων 15, και μόνο 20% στι 12 χώρε μέλη μετά τη διεύρυνση. Και αυτό με βάση τα στοιχεία του 2007 που μας δίνει η Eurostat. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που είναι γνωστό, αλλά που ίσως δεν έτυχε της δέουσας προσοχής μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχει εναλλαγή, δεν υπάρχει αντικατάσταση. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που να λαμβάνουν τη σκητάλη από τους παλιότερους γεωργούς. Γιατί οι, πιο ηλικιωμένοι γεωργοί συνεχίζουν την γεωργική τους δραστηριότητα και μετά το όριο συνταξιοδότης στα 65 χρόνια. Γιατί δεν υπάρχουν αντικαταστάτες. Για ποιους λόγους, ποια είναι τα βασικά αίτια Πώς εξηγείται αυτή η έλλειψη ενδιαφέροντος, αυτή η αδιαφορία των νέων για ανάληψη γεωργικής δραστηριότητας. Τα αίτια μπορεί να είναι πολλά και διάφορα. Υπάρχουν όμως ε, κάποιες κοινωνικές και οικονομικές αιτίες. Και αν αστιαστούμε σε αυτές, διαπιστώνουμε ότι έχουμε τρία βασικά στοιχεία που είναι αποτρεπτικά για τους νέους. Και αναχαιτίζουν ή παρεμποδίζουν και την, ε, τους νέους από την ε, ενασχόληση με τη γεωργία. Ο πρώτος παράγοντας από τους τρεις που είναι φάμιλοι στο βάρος τους και μάλιστα έχουν ε, μια συμπληρωματικότητα μεταξύ τους αυτοί οι τρεις παράγοντες. Ο βασικός παράγοντας, ο πρώτος παράγοντας είναι η, η δυσκολία να έχει κανείς μια βιώσιμη γεωργική εκμετάλλευση. Δηλαδή να μπορεί να έχει μια οικονομική βιωσιμότητα. Στο κείμενο που έχετε υπάρχει ένας ορισμός της βιωσιμότητας. Ουσιαστικά μιλούμε για τη δημιουργία μιας γεωργικής εκμετάλλευσης που θα έχει τουλάχιστον 40 μονάδες ε, οικονομικής διάστασης ε, ώστε να εξασφαλίζει μια ελάχιστη βιωσιμότητα. Και όταν βλέπουμε τα χαρακτηριστικά της πλειοψηφίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση τις οικονομικές διαστάσεις, βλέπουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων πόρο απέχει από το όριο της βιωσιμότητας. Οπότε είναι προφανές ότι δεν είναι και πολύ ελκυστικό για ένα νέο να ξεκινήσει μια τέτοια δραστηριότητα, διαπιστώνοντα ότι δεν είναι εξασφαλισμένη ε, η βιωσιμότητα και ο βιοπορισμό. Οπότε, γιατί να εμπλέκει σε αυτή τη διαδικασία ο νέο. Μία συναφή αιτία είναι και μια κοινωνική αιτία που σχετίζεται με την απασχόληση. Οι επαγγελματίες ε, νέοι γεωργοί θα μπορούσαν να αναλάβουν ε, μια γεωργική εκμετάλλευση, είχαν τουλάχιστον μια μονάδα εργασίας ετήσια. Ενώ τα ποσοστά που περιλαμβάνει η έκθεση δείχνουν ότι ναι, με στι 15 χώρες Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπερνούμε αυτό το λόγο κατά μέσο όρο για όλε τι 15 ε, παλιέ χώρες Ευρωπαϊκή Ένωση, στι νέε 12 χώρες Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε πολλέ ε, γεωργικές εκμεταλλεύσει ε, που εξασφαλίζουν έστω και μία θέση απασχόληση, μία μονάδα απασχόληση ετησίω στο γεωργό. Εξού και η δυσκολία δημιουργία θέσεων απασχόληση, για του νέου που θα ασχοληθούν με τη γεωργία η γεωργία δεν είναι ελκυστική εξαιτία αυτών των παραγόντων. Και υπάρχει ένα τρίτο στοιχείο, ένα τρίτο παράγοντα, που είναι επίση αποφασιστική σημασία, γιατί επαναλαμβάνω είναι εισάξει σε βάρο, εφάμιλη σε βάρο οι τρει παράγοντε. Είναι ότι είναι δύσκολο με τη γεωργική ε, δραστηριότητα να επιτύχει κανεί ένα επίπεδο εισοδήματο που να επιτρέπει το βιοπορισμό από τη γεωργία. Και από αυτή την άποψη είναι χαρακτηριστικό ότι η κοινή γεωργική πολιτική σχετίζεται άμεσα με αυτή τη δυνατότητα εξασφάλιση ενός ε, ικανοποιητικού εισοδήματο. Γιατί σε αυτό το εισόδημα περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις. Και οι ενισχύσεις με βάση και εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, που πέρασε και από την Επιτροπή σας, διαπιστώνεται ότι οι ενισχύσεις έχουν αποκτήσει όλο και μεγαλύτερο βάρος στο συνολικό εισόδημα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ιδιαίτερα στις ε, μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Οπότε, το κατά πόσο κανείς έχει πρόσβαση ή όχι στο καθεστώς της ενίσχυσης, στις άμεσες ενισχύσεις, είναι μια πολύ σημαντική προϋπόθεση για να ενταχθεί ένας νέος στο επάγγελμα. Αν ένας νέος δεν έχει το εχέγγυο ότι θα έχει πρόσβαση σε τέτοιες ενισχύσεις, πολύ δύσκολα θα στραφεί προς τη Γεωργία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πολύ μεγάλο διάστημα και η κοινή γεωργική πολιτική γενικώ εφάρμοσε κάποια μέτρα για να βελτιώσει την κατάσταση και πολιτικές. Και οι πολιτικές είχαν κάποια αποτελέσματα. Οι πολιτικές ε, είναι απλές. Ήταν κυρίως τρεις οι δρόμοι για να γίνει κανείς ε, γεωργός. Να κληρονομήσει μια γεωργική εκμετάλλευση, να παραλάβει από κάποιον πρόωρο συνταξιοδοτούμενο ή να μπει νέος γεωργός. Αυτή ήταν οι τρεις διαβλή εισόδου στη γεωργία. Το πιο δύσκολο βέβαια είναι να, είναι, να γίνει κανείς γεωργός χωρίς να έχει προηγούμενα κληρονομήσιμη εκμετάλλευση να διαδεχθεί κάποιον. Και οι πολιτικές ήταν τέσσερις ανάλογα με τις διάβλους και ανάλογα με τη διάβλο είχαμε και διαφορετικές πολιτικές. Ό,τι αφορά την κληρονομιά έχουμε πολύ λιγότερες ε, πολιτικές γιατί όποιος κληρονομεί την γεωργική εκμετάλλευση κληρονομεί και την πρόσβαση στο καθεστώς ενίσχυσης. Οπότε την ε, πρόσβαση στην ενίσχυση την έχει, το α το έχει. Τώρα χρειάζεται το ΣΕ, δηλαδή κάποιες ενισχύσεις επενδυτικές, για να μπορέσει να βελτιώσει με επενδύσει την γεωργική του εκμετάλλευση. Τώρα, η δεύτερη διάβλος, μέσω της πρόορισης συνταξιοδότησης. Εκεί είχαμε τα μέτρα B, ε, C και D. Είναι σημαντικά αυτά τα μέτρα, το BCD, γιατί εκεί έχουμε την ενίσχυση για να ενθαρρύνουμε τους νέους, για τον κύριο νέοι, τους νέους γεωργούς για να τους ελκύσουμε με, το, με, αυτό, αυτή την επιδότηση ε, της ε, έναρξης της νέας επιχειρήσης, το Startup Aid. Επίσης, ε, ενισχύσεις για τις επενδύσεις και ε, το ΔΕΛΤΑ είναι η ενίσχυση προς αυτόν που συνταξιδοτούνταν πρόδρα. Και η εξνόβο, η τρίτη κατηγορία, είχαν ε, μέτρα και από τις τρεις πολιτικές, α, β και γ. Στους νέους γεωργούς ε, δίνονταν η ευκαιρία από τα εθνικά αποθεματικά να αποκτήσουν κάποια συγκεκριμένα δικαιώματα. Βέβαια, τα υποθεματικά αυτά δεν λειτουργήσαν και πολύ καλά, οπότε δεν δόθηκαν εγγυήσει για τα δικαιώματα αυτά στους νέους Γιώργους, Ούτε και τα πολύ μεγάλα τα ποσά στα αποθεματικά αυτά. Πώς μπορούμε να συνοψίσουμε τα αποτελέσματα από το καθεστώ νέων γεωργών. Τα αποτελέσματα ήταν δυστυχώ ελάχιστα για την προσέλκυση νέων γεωργών. Η εμβέλεια των νέων μέτρων και τα κίνητρα που δόθηκαν ήταν ανεπαρκή. Έτσι είχαμε ελάχιστη ανάληψη δραστηριοτήτων από νέους. Είχαμε τρει, άντε, περίπου χιλιάδες νέους ε, γεωργούς για μία τετραετία. Βλέπετε πόσο πενιχρά είναι αυτά τα στοιχεία, πόσο αμεληταία. Τα μέτρα εξυγχρονισμού που δεν κάνουν διακρίση μεταξύ νέων και πιο ηλικιωμένων γεωργών, γιατί είναι μικτές ε, για τις εκμεταλλεύσεις. Αυτά τα μέτρα ήταν πολύ πιο χρήσιμα και σίγουρα ένα τμήμα αφορούσαν τους νέους γεωργούς, προβλέποντας και ένα ε, σχέδιο εξυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Αυτά ήταν γύρω σε 100.000. Και ένα μέτρο που δεν είχε και μεγάλη επιτυχία ήταν αυτό της πρόορης συνταξιοδότησης. 19.000 δικαιούχοι μόνο για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα σε μία τετραετία. Διαπιστώνεται ότι το αποτέλεσμα αυτό είναι αμεληταίο. Και μάλιστα σε ορισμένε χώρε, στι χώρε ε, μετά τη διεύρυνση, μόνο η Πολωνία έχει το 80% αυτών των αποτελεσμάτων, μία και μόνο χώρα. Οπότε, τι γίνεται. Η κατάσταση είναι σχετικά εύθραυστη, η πολιτική είναι ανεπαρκής και ελάχιστα κίνητρα δίνει στους νέους γεωργούς για να αναλάβουν ε, γεωργικές δραστηριότητες. Οπότε οι νέοι δεν ε, βρίσκουν ελκυστικές προϋποθέσεις για να ασχοληθούν με τη γεωργία, αλλά και οι γεωργοί δεν ε, βρίσκουν αρκετά κίνητρα για να εγκαταλείψουν τη γεωργία προτιμούν να συνεχίσουν την δραστηριότητά του στη γεωργική παρά να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα. Γιατί δεν υπάρχουν αρκετά μέτρα που να ενθαρρύνουν και την πρόωρη συνταξιοδότηση. Έχουμε τώρα και μια νέα πρόταση που τη γνωρίζετε, πρόταση των νέων κανονισμών που υπόκειται φυσικά σε αναθεωρήσεις. Ο κύριος Καπόλα Σάντος ασχολήθηκε με τους κανονισμούς αυτούς ε, στις εκθέσεις του, τις μελετήσαμε πολύ σχολαστικά και υπάρχει κάποια βελτίωση σχέση με την παρούσα κατάσταση. Το μοντέλο είναι το ίδιο, αλλά ενισχύεται κάπως. Βλέπετε με πορτοκαλί τα μέτρα που ενισχύονται, Το μέτρο α, δηλαδή πρόσβαση στο καθεστώς ενίσχυσης. Πολύ σημαντικό μέτρο για να εξασφαλιστεί το γεωργικό εισόδημα. Τώρα θα έχουμε ένα νέο μέτρο, ένα συμπληρωματικό ε, επίδομα, καλύτερη λοιπόν ε, ενίσχυση, βελτιωμένη ενίσχυση για τους νέου για τους νέους γεωργούς που θέλουν να εισέλθουν στο επάγγελμα. Αυτό συζητάται μεταξύ άλλων με τους νέους κανονισμούς. Επίσης και το μέτρο Β, ε, βοήθεια για νέα επιχείρηση, το startup. Και αυτό το μέτρο βελτιώνεται με ένα νέο σύστημα καλύτερης αξιολόγησης ε, ε, των εκμεταλλεύσεων και το μέτρο επίσης ενισχύεται με ένα σύστημα βελτίωσης της ε, χρηματοδότησης των ε, επιχειρηματικών σχεδίων που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να έχει κανείς δικαίωμα ε, για την ενίσχυση. Και εμφανίζεται και μία, ένα νέο μέτρο που αντικαθιστά το προηγούμενο εξαφανίζεται η πρόορη συνταξιοδότηση και εμφανίζεται το Small Farmer Scheme, το καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές, που δίνει μια δυνατότητα πρόορης ε, συνταξιοδότησης. Γιατί δίνεται ένα πριμ σε αυτόν που εγκαταλείπει την μικροκαλλιέργεια. Αλλά αυτό το μέτρο δεν ε, ε, προτάθηκε για την πρόορη συνταξιοδότηση, αλλά για να ξεκονομηθούν κάποια κονδύλια κυρίως από τις ενισχύσεις για τις μικροκαλλιέργειες και βλέπετε στην έκθεση τονίζουμε αυτό το σημείο. Φαίνεται όμως ότι και η νέα πρόταση δεν είναι επαρκής. Παρόλο που έχει κάποιες ε, δυνατότητες βελτίωσης. Οι άμεσες πληρωμές, οι άμεσες ενισχύσεις από τα εθνικά αποθεματικά βελτιώθηκαν μεν, αλλά δεν είναι πολύ εντυπωσιακή βελτίωση. Επίσης, ε, η διεύρυνση του, ε, της επιχορήγησης με την προϋπόθεση του επιχειρηματικού σχεδίου είναι σωστή, αλλά δεν είναι αποφασιστική σημασία. Ουσιαστικά προϋπήρχε λιγότερο ή περισσότερο υποχρεωτική. Τώρα δίνεται μια προθεσμία, εξάμεινη προθεσμία για να διεκπαιρεωθεί αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο. Επίσης, η επενδυτική υποστήριξη και αυτό το μέτρο υπήρχε, τώρα ενισχύεται με ένα άλλο σημαντικό θέμα που γίνεται πιο ρητό, που είναι το θέμα της υποστήριξης ε, της γης. Το θέμα της γης είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα δικαιώματα πληρωμής ε, συνδέονται με, την, ε, με τη γη για να έχει κανείς δικαίωμα στην ενίσχυση. Και υπάρχει όμως μια σημαντική στενοπός που τονίζεται. Το θέμα είναι να υπάρχουν αρκετά δικαιώματα ενίσχυσης και φυσικά και αρκετές γέες για να μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση. Και υπάρχει και το περίφημο νέο καθεστώς για τις μικροκαλλιεργητές που όπως είπα και προηγουμένως ε, από μόνο του δεν πρόκειται να ελκύσει πολλούς νέους γεωργούς στο επάγγελμα. Δεν είναι ούτε ο στρατηγικός στόχος ούτε το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Οπότε Συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι ανεπαρκής, είναι ατελής. Αυτό είναι το πόρισμα αυτής της ανάλυσης. Για ένα νέο Γιώργο. Ας πάρουμε μια ακραία περίπτωση. Τον εξνόβο που δεν έχει ούτε κληρονομήσει ούτε διαδεχθεί κάποιον προώρα εξοδοτούμενο. Γιατί σκεφτόμαστε ότι μπορούν από κάποιοι άνεργοι να θελήσουν να ασχοληθούν με τη γεωργία. Έχασαν τη δουλειά τους κάπου αλλού, να αποφασίσουν ξαφνικά να ασχοληθούν με την γεωργία λόγω της κρίσης. Αυτή είναι η εξνόβο. Για αυτούς ε, ε, το θέμα της ενίσχυσης, της άμεσης ενίσχυσης θα είναι τεράστια στενοπός και θα αναχαιτήσει τους νέους αυτούς γεωργούς. Δεύτερο στοιχείο. Η επιχορήγηση που είναι μέχρι, και, μέχρι 70.000 ευρώ μετά το διαγνωστικό έλεγχο, το health check ε, ανέβηκε από 50 σε 70 χιλιάδες. Τελικά ο μέσος όρος είναι γύρω στους 40.000 χιλιάδες. Δεν πρόκειται να ανεβεί ποτέ στα 70.000 χιλιάδες γιατί ε, υπάρχει συγχρηματοδότηση, οι χώρες έχουν κρίση οπότε δεν ε, ε, μπορούν να μεγαλώσουν αυτό το ποσό. Εν πάση περιπτώσει, 40-42 χιλιάδες ευρώ για ένα νέο δεν είναι επαρκέ κίνητρο ή έναυσμα για να λάβει την απόφαση να μπει στη Γεωργία όταν ξέρετε δεν υπάρχει βιοπορισμός εξασφαλισμένος και δεν υπάρχει καμία εγγύηση για επαρκέ εισόδημα εφόσον δεν έχει εξασφαλισμένα δικαιώματα ενίσχυση. Οπότε δεν νομίζω να λειτουργήσει και πολύ το μέτρο. Το θέμα του εξυγχρονισμού. Μέχρι στιγμής έχει λειτουργήσει αρκετά καλά, θα πρέπει να ενισχυθεί. Και μάλιστα υπάρχουν στοιχεία ε, για κάποιε χώρε που δείχνουν ότι οι περικοπέ αφαιρούν κονδύλια από τον εξυγχρονισμό. Γιατί ο δεύτερο πυλώνα τη ΠΑΚΟ, ο εξυγχρονισμό, απορροφά πάνω από το 10%. Οπότε εκεί υπάρχουν κονδύλια για περικοπέ. Αλλά το, τα προγράμματα για του νέου είναι 3% και δεν υπάρχουν κονδύλια για περικοπέ. Οπότε το πιο ισχυρό μέτρο του εξυγχρονισμού είναι αυτό που θα υποστεί τι περισσότερε περικοπέ και άρα θα αποδυναμωθεί. Γιατί εκεί υπάρχουν κονδύλια, από εκεί θα κόψουν. Και τέλο υπάρχει και το τελευταίο μέτρο, το Small Farmer Scheme, αυτό το μέτρο για του μικροκαλλιεργητέ. Εκεί δεν περιμένουμε και πολλά αποτελέσματα, εντυπωσιακά τουλάχιστον. Οπότε οδηγούμε στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να τη διευρύνουμε και ίσως να υιοθετήσουμε και μια νέα προσέγγιση, μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση. Γιατί το κείμενο μιλά για συμπληρωματική πρόταση. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Θέλουμε να οικοδομήσουμε, να φτιάξουμε, όχι να αρνηθούμε, να καταστρέψουμε. Θέλουμε να βελτιώσουμε τα υπάρχοντα. Οπότε καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα που είναι και το πιο καινοτόμο στοιχείο της έκθεσης. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ε, έλλειψης των νέων γεωργών. Θα μπορούσαμε αυτό το πρόβλημα να το θεωρήσουμε όχι ως τομεακό πρόβλημα, κλαδικό της γεωργίας, αλλά ως ε, εδαφικό πρόβλημα, πρόβλημα της υπαίθρου, γεωγραφικό. Αυτό δεν είναι κάτι τελείως ε, το έχουμε ακούσει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν σχολιαστεί παρόμοιες προσεγγίσεις. Αλλά για το συγκεκριμένο θέμα θα προσπαθήσω να το συγκεκριμενοποιήσω. Θεωρώ ότι η εδαφική, η γεωργική προοπτική θα δώσει μια νέα όθηση προκειμένου να καλυφθεί αυτό το οξύ πρόβλημα της έλλειψης νέων γεωργών. Και αναλύοντας τα αίτια αυτού του φαινομένου, θα ήθελα να λάβουμε υπόψη και ένα τέταρτο παράγοντα, ένα τέταρτο αίτιο, που είναι πάνω από τους ε, τρεις ε, παράγοντες που είναι πιο τομεακοί αφορούν μόνο τη γεωργία. Αυτός ο τέταρτος παράγοντας αφορά την παρούσα κατάσταση του γεωργικού κλάδου και της υπαίθρου στις, ε, στις ζώνες που δεν έχουμε νέους γεωργούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί για να αναλάβει κανείς μια γεωργική δραστηριότητα δεν χρειάζεται μόνο να βρει ένα τομέα που θα είναι εύκολη η είσοδός του, να έχει ένα επίπεδο βιωσιμότητας, να εξασφαλίζει βιοπορισμό και εισόδημα. Θα πρέπει να δει αν το συνολικό περιβάλλον είναι πρόσφορο για να ασχοληθεί κανείς με μια γεωργική δραστηριότητα. Γιατί ε, από ό,τι φαίνεται ο Γιώργος δεν θα μπορέσει να ζήσει μόνο από τη γεωργία. Οι περισσότεροι γεωργοί είναι μερικής απασχόλησης γεωργοί. Οπότε από τη στιγμή που είμαι καταδικασμένο σε μερική απασχόληση, για να ασχοληθώ με τη γεωργία, θα προσπαθήσω να βρω ένα περιβάλλον που θα μου επιτρέπει και άλλε διεξόδου. Οπότε, ο εδαφικό αυτό παράγοντα του συνολικού περιβάλλοντο θα πρέπει να προσθεθεί στου προηγούμενου τρει που έχουν αμυγή σύνδεση με τη γεωργία, με τον ίδιο τον κλάδο. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν ποια θα πρέπει να είναι τα νέα μέτρα και ίσως ε, δεν θα έχουμε μόνο ένα απλό μοντέλο για τη συμπερίληψη νέων ή λιγότερο νέων στη Γεωργία, να περάσουμε σε ένα νέο ε, για το κατά πόσο ε, θα μπορούσε κανείς κάποιος να εγκατασταθεί σε, στην Ήπεθρο, σε ένα περιβάλλον αγροτικό. Το θέμα δεν είναι πόσοι είναι γεωργοί. Το θέμα είναι ότι στις περισσότερες αγροτικές ζώνες υπάρχουν ελάχιστοι κάτοικοι και κυρίως ελάχιστοι νέοι που θα ασχοληθούν με οποιοδήποτε επάγγελμα στην Ήπεθρο. Οπότε εκεί έχουμε ένα νέο καθεστώς όπου η διεύλη εισόδου στην οικονομική δραστηριότητα στις αγροτικές περιοχές και στην Ήπεθρο θα ήταν δύο. Ή θα μπει κανείς ως επαγγελματίας γεωργός, νέος γεωργός, ή ως νέος ή λιγότερο νέος ε, ενεργός στο γεωργικό κλάδο. Δεν είναι ασύμβατα αυτά τα δύο θέματα, γιατί μπορεί κανείς να είναι, να είναι μερική απασχόληση νέος γεωργό ή από την άλλη να ενεργοποιείται κάπου στην Ήπεθρο. Ή άλλος μπορεί να είναι αποκλειστικά και μόνο γεωργός ή ε, να έχει μία δραστηριότητα στην Ήπεθρο. Ω νέος γεωργός ε, μπορεί να υποφεληθεί από τα τέσσερα μέτρα που είπαμε και τις νέες προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΑΒ, Γ και Δ. Και με τις βελτιωμένες φυσικά προτάσεις που σας παρουσίασα. Αν μπω, μπω όμως ως νέος γεωργός μερικής απασχόλησης ή νέος ή λιγότερο νέος, νέος γεωργός μερικής απασχόλησης ή που θα δραστηριοποιούμε στην, στην Ήπεθρο, σε τέτοια περίπτωση χρειάζομαι και άλλα μέτρα για να μπορέσω να εγκατασταθώ σε ένα αγροτικό περιβάλλον στην Ήπεθρο. Εκεί δεν, χρειά, αρκεί η γεωργία. Πρέπει να έχω και άλλες διεξόδους επαγγελματικές. Στην Ήπεθρο μεν, αλλά διέξοδο πέρα από τη γεωργία. Και εκεί προτείνω τέσσερα νέα μέτρα που δεν περιλαμβάνονται στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά εμέσως ε, υπονοούνται σε διάφορα άλλα σημεία της πρότασης. Και παραλαμβάνω, το σύστημα προτείνω είναι συμπληρωματικό, δεν είναι εναλλακτικό. Και σας αναφέρω τέσσερα μέτρα. Το πρώτο είναι πολύ σημαντικό γιατί ουσιαστικά Μα προτείνει ένα εισόδημα για του νέου. Νομίζω ότι αυτό το μέτρο θα μπορούσαμε να το δεχτούμε. Και από τη στιγμή που επιδοτούμε ένα νέο γεωργό για να ενταχθεί με ένα πριμ νέα επιχείρηση, γιατί να μην δώσουμε και μια επιχορήγηση σε έναν νέο ε, προσωρινά για να παραμείνει στην Ήπεθρο, έστω και αν είναι μερικής απασχόλησης Γεωργός. Τώρα, πόσο, σε τι να ανέρχεται αυτό το πριμ, να είναι το ίδιο με αυτό που δίνουμε στο νέο γεωργό, τουλάχιστον. Αλλιώ θα έρθω σε διακριτική μεταχείριση. Αν θέλω να, γίνω νέο γεωργό, έχω ε, πριν. Αν όμω θέλω να ασχοληθώ με μια δραστηριότητα αγροτική, δεν την έχω, είμαι μια δραστηριότητα στην Ήπεθρο. Γιατί όχι. Ένα άλλο μέτρο που υπάρχει, αλλά είναι πολύ ασθενές και καλό θα ήταν να ενισχυθεί. Είναι γνωστό αυτό το μέτρο, και αφορά τα μέτρα της μεθόδου Leader. Όσοι παρακολουθήσαμε, μπήκαμε στον κόπο να παρακολουθήσουμε τα χρόνια αυτά το πρόγραμμα Leader, διαπιστώσαμε ότι ήταν πολύ επιτυχημένο και ταυτόχρονα και αποτυχημένο. Η μέθοδος Leader είναι μια μέθοδος σημαντικής επιτυχίας. Όλοι το δέχονται και συμφωνούν. Και είχε πολύ σημαντικό αντίκτυπο, πολύ μεγάλη απήχηση παρόλα αυτά δεν αξιοποίησε πλήρως το δυναμικό του αυτό το πρόγραμμα Leader. Και στον κανονισμό βλέπουμε ότι προβλέπεται τουλάχιστον 5% για το Leader. Είναι ανεπαρκές αυτό το ποσό. Θα παραμείνει περιθωριακό αυτό το πρόγραμμα. Και θα ξέρετε ότι το τελευταίο καιρό το Leader δεν καλύπτει καν ε, τις ε, δεσμεύσεις ε, υποχρεώσεων, γιατί υπάρχουν προβλήματα στη συγχρηματοδότηση, αλλά υπάρχουν και προβλήματα χρηματοδότησης των, επιχειρηματικών σχεδίων. Από πού θα βρεθούν κονδύλια για τα νέα επιχειρηματικά σχέδια, ποιος θα δώσει πιστώσεις. Οπότε εκεί θα είχαμε ένα σημαντικό μέτρο αν ενισχυθεί. Φυσικά το αστέρι αυτών των προτάσεων, κορονίδα αυτών των προτάσεων που ε, λέμε πολιτική για την ύπεθρο εντός της ΚΑΠ και του δεύτερου πυλώνα. Κατά τη γνώμη μου, η κορονίδα των μέτρων είναι το μέτρο ΣΕ, το μέτρο Γ. Community-led support, δηλαδή εφαρμογή κατά κάποιο τρόπο της μεθόδου του leader με την ε, ταυτόχρονη εφαρμογή όλων των ταμείων σε, ε, σε μια συγκεκριμένη περιοχή του ΦΕΝΤΕΡ, του Κοινωνικού Ταμείου και του ΦΕΝΤΕΡ. Θα έχουμε συρροή όλων των κονδύλιων των τριών ταμείων σε συγκεκριμένη περιοχή. Και από ενοιολογική άποψη αυτό το μέτρο θα ήταν πολύ πετυχημένο. Βέβαια, διαβάζοντας τον κανονισμό που αφορά αυτά τα μέτρα, αν είχατε την ευκαιρία να ρίξετε μια ματιά, διαπιστώνετε ότι είναι τόσο περίπλοκη η διατύπωση και τόσο δύσχερη ο κανονισμός και τόσο περίπλοκη η γραφειοκρατία που τον κάνει πραγματικά δυσεφάρμοστο και δύσχριστο. Οπότε η επιτυχία είναι μάλλον θεωρητική παρά πρακτική. Υπάρχει όμως η δυνατότητα. Αλλά είναι κρίμα να αποκλίνουν τα διάφορα ταμεία, να πηγαίνει προς τη μία το κοινωνικό ταμείο, προς την άλλη το ΦΕΝΤΕΡ και προς την τρίτη κατεύθυνση το ΦΕΑΝΤΕΡ. Γιατί το 99 θα θυμάστε, είχαμε τις ζώνες 5Β. Για τις ζώνες 5Β είχαμε ε, ολοκληρωμένη πολιτική για την Ήπεθρο. Γιατί να μην ε, επανέλθουμε σε μια ολοκληρωμένη πολιτική για την Ήπεθρο που είχαμε το 99. Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό, με, με το συνδυασμό των ταμείων, θα έχουμε μια πολύ καλύτερη ολοκλήρωση. Τότε είχαμε τις περιοχές βέβαια τύπου 2, τις ε, ανεπτυγμένες, όχι τις περιοχές του στόχου 1. Και αυτή ήταν η βασική δυναμία του μέτρου τότε το 1999. Πάντως το μέτρο αυτό δεν είναι καινούργιο, θα μπορούσαμε να το ανακτήσουμε και να το αξιοποιήσουμε. Και υπάρχουν κάποια μέτρα που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά στις αρμοδιότητες των χωρών. Είναι τα μέτρα H, ETA, που είναι εθνικές πολιτικές, αφορούν τις εθνικές πολιτικές. Η πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως ε, των πρώτων βασικών χωρών έχουν, όλες οι χώρες έχουν τις δικές τους πολιτικές αγροτικές και τις υπαίθρου που χρησιμοδοτούν με τους δικούς τους κανονισμούς. Αυτές οι πολιτικές καλό θα ήταν να συγκλίνουν σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο και να γίνονται πιο συναφείς μεταξύ τους. Οπότε φτάνουμε τώρα και ολοκληρώνω εδώ σε αυτό που ζητούμε για να δοθούν ενάυσματα για τους νέους γεωργούς. Και νομίζω ότι είναι πολύ συγκροτημένο το συμπέρασμα. Θέλουμε όχι μόνο να ενισχύσουμε τα υφιστάμενα μέτρα που είχαν μέχρι στιγμή με μικρότερη ή μεγαλύτερη επιτυχία. Αυτό που ζητούμε είναι να έχουμε μια πραγματικά ε, ευρωπαϊκή πολιτική για την Ήπεθρο. Μόνο μια τέτοια πανευρωπαϊκή πολιτική για την Ήπεθρο θα μπορέσουμε να στηρίξουμε την είσοδο των νέων γεωργών και των νέων εργαζόμενων στην Ήπεθρο. Γιατί η θεμελιώδη πρόκληση για τα επόμενα χρόνια θα είναι η σπάνιση των νέων γεωργών. Αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε έλλειψη και νέων επιχειρηματιών στη, στην Ήπεθρο. Νέων ή λιγότερο νέων. Γιατί είναι αλήθεια ότι η λιγοτερων νεων γιατι ειναι αληθεια οτι η γεωργια σε μερική επασχόληση είναι το, το κανόνας πια στις περισσότερες χώρες. Και αυτό είναι γεγονός. Οπότε από τη στιγμή που είναι γεγονό η μερική απασχόληση στη Γεωργία, αποδεχτούμε ότι δεν είναι επαγγελματίε αυτοί οι Γεωργοί. Να μην επικεντρώνουμε μόνο τα μέτρα στου επαγγελματίε Γεωργίου. Δεν λέω ότι δεν θα πρέπει να ε, επιδοτήσουμε του επαγγελματίε Γεωργού, αλλά να μην ξεχνούμε και του υπόλοιπου Γεωργού, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία, που είναι μερική απασχόληση Γεωργοί. Το 80% είναι κάτω των 40% ε, και 90% ε, είναι στις νέες χώρες ε, της τελευταίας διεύρυνσης. Οπότε είναι μεγάλος ο αριθμός αυτών των μερικής απασχόλησης γεωργών. Και τέλος, ε, η σημασία του εδάφους της περιοχής γενικώ. Το έδαφος είναι πολύ σημαντικός παράγοντας και αμελήθηκε στις κοινοτικές πολιτικές, ιδιαίτερα στην κοινή γεωργική πολιτική. Σίγουρα έχουμε ζώνες, έχουμε περιοχές, έχουμε ε, μειονεκτούσες περιοχές, είχαμε την περιφερειακή πολιτική, τις διάφορες κατηγορίες περιφερειών, έχουμε ζώνες ειδικού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, ζώνες με διάφορα προτερήματα, αλλά δεν έχουμε πραγματικά πολιτικές ανά ε, εδαφική μονάδα. ΝΑΤ 4. Υποπεριφερειακές ζώνες έχουν στατιστική αξία, αλλά δεν έχουν πολιτική αξία αυτές οι ζώνες ό,τι αφορά την εφαρμογή των πολιτικών. Χρειαζόμαστε υποπεριφερειακές, υποεπαρχιακές ζώνες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οπότε θα θέλαμε να ζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Πολιτική να βάλει μια τάξη σε όλα αυτά, προτείνοντας μια νέα πολιτική για την Ήπεθρο και που θα περιλαμβάνει όλα αυτά τα μέτρα που ισχύουν. Αυτό είναι ο πίνακας πολύ απλός και τελειώνω με αυτό. Χρειαζόμαστε μια νέα πολιτική για την Ήπεθρο που θα περιλαμβάνει τα μέτρα τη κοινή γεωρική πολιτική. Αυτά που σχολιάσαμε προηγουμένω. Τα βελτιωμένα μέτρα όμω. Επίση, χρειαζόμαστε μια πολιτική για την Ήπεθρο που θα ε, περιλαμβάνει και κάποιε πολιτικέ συνοχή για την Ήπεθρο. Χρειαζόμαστε μια πολιτική για την Ήπεθρο που θα δίνει νόημα στι εθνικέ πολιτικέ. Δεν θέλω να μιλήσω για άλλε χώρε, αλλά υπάρχουν χώρες που εφαρμόζουν πολύ πιο ισχυρές πολιτικές για την Ήπεθρο από ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν παράδοση και έχουν ε, πολύ σημαντικές νομοθεσίες και πολύ σημαντικούς προϋπολογισμούς για την Ήπεθρό τους. Οι πολιτικές αυτές λοιπόν θα πρέπει να σειραίουν προς ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα τους δίνει νόημα. Και αυτό είναι το νέο καθεστώς της ευρωπαϊκής πολιτικής για την Ήπεθρο. Αν τα κάνουμε όλα αυτά, να είστε βέβαιοι ότι θα βελτιώσουμε και την, παρουσίαση των, την παρουσία των γεωργών και κυρίως την παρουσία νέων γεωργών και νέων ε, απασχολούμενων στην Ήπεθρο γενικό. Έχουμε πολλά στοιχεία, έχουμε πολλούς πίνακες στην έκθεση και στη μελέτη. Αν έχετε χρόνο, ρίξτε μια ματιά στην οριστική έκθεση και είμαι στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε απορίες και συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε καθηγητά κύριε Γκονζάλες για την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη σας. Ξεκινάμε τώρα τη συζήτηση. Έχουν ζητήσει το λόγο ο Αντίπροεδρος Μποβέ. Ξεκινάμε με τον Ζωζεφ. Oui, euh, Ναι. Άκουσα την παρουσίασή σας. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία νομίζω ότι δεν ε, ε, υπάρχουν ή τουλάχιστον δεν μπορεί να βρει κανείς στατιστικά, ότι δηλαδή πολλές χώρες ε, υπάρχουν όπου οι πραγματικές ε, εγκατεστημένες ε, ανάγκες ε, είναι ίσες με τους γεωργούς οι οποίοι βοηθούνται. Το βλέπουμε και στη Γαλλία. Δηλαδή υπάρχει ένας διπλασιασμός των εγκαταστάσεων. Πώς μπορούμε λοιπόν να δείξουμε ότι η ενίσχυση δεν είναι προσαρμοσμένη τουλάχιστον για το ίμιση των ατόμων. Επίσης αναφερθήκατε στην πρόσβαση στη γη. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπάρχει εθνική μάλλον ευρωπαϊκή νομοθεσία. Διαφέρουν οι νομοθεσίες κατά χώρα και μάλιστα πάρα πολύ. Και για μένα αυτό είναι ένα από τα βασικά προβλήματα, δηλαδή η πρόσβαση στη γη είτε ιδιόκτητη είτε νοικιασμένη, πώς θα γίνει μια ε, πολιτική προσβάσεω στη γη για την ε, ε, πρόσβαση και για την μεταβίβαση. Επίσης η μεταβίβαση είναι μία τροχοπέδη που αντιμετωπίζουμε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή το χαμηλό επίπεδο των ε, γεωργικών συντάξεων. Δηλαδή οι συντάξεις είναι πολύ χαμηλές και ως εκ τούτου παρατείνει κανείς την γεωργική δραστηριότητα γιατί ε, συνεχίζονται οι ενισχύσεις και ο όγκος είναι μεγαλύτερος από τη ε, σύνταξη. Και αυτό είναι το δεύτερο πρόβλημα. Και το τρίτο που είναι πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι τα, τα, τα μοντέλα, δηλαδή οι, τα αγροκτήματα που μεταβιβάζονται ε, γίνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε είναι δύσκολο να αναλυφθούν από τους νέους. Χρειάζονται τόσα χρήματα ώστε δεν πρόκειται να αποδώσουν το αντίστοιχο εισόδημα. Ε, αυτό λοιπόν το καπιταλιστικό είδος εκμεταλλεύσεως είναι βιώσιμο για την επόμενη γενιά. Και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να θέσουμε γιατί βλέπουμε μεγάλες εγκαταστάσεις που δεν βρίσκουν αγοραστή στη συνέχεια. Αυτό ήθελα να σας ε, κάνω, αυτές τις τρεις ερωτήσεις. Ευχαριστώ Ζωζέ. Τώρα ο Αλμπερντές και μετά ο κύριος Άγνιου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για τις πληροφορίες. Οι πληροφορίες σας όμως με επιβεβαιώνουν την άποψή μου ότι από την ε, Βρυξέλλες δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα της Ευρώπης. Είναι πολύ πιο πολυσχηδής η Ευρώπη και δεν μπορούν οι Βρυξέλλες ε, να υπαγορεύσουν τους όρους. Εδώ και στην ε, Γερμανία διαφέρουν οι όροι. Εγώ είμαι από τη Βαβαρία και βλέπω ότι οι νέοι τσακώνονται για κάθε εκτάριο το οποίο ενοικιάζεται και εάν ε, ρυθμίσουμε τα θέματα από τις Βρυξέλλες θα ανεβούν ε, τα νίκια εκμεταλλεύσεως. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε όλα αυτά να τα εκτονώσουμε διότι βλέπουμε ότι υπάρχει τέτοιος ανταγωνισμός ώστε δεν υπάρχει επαρκής γη προς εκμετάλλευση και όταν αν δεχθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόταση Τσόλος, του Επιτρόπου δηλαδή, ε, θα ανέβει πάλι 200, κατά 200 ευρώ το τίμημα για το ένα εκτάριο και θα έχουμε και άλλα προβλήματα. Πρέπει να κάνουμε στοχευμένες ε, δράσεις. Δεν θέλω να μιλήσω για την ΤΕΓΕΜΠΕ που αντιμετωπίζει προβλήματα, αλλά δεν μπορούμε εμείς να λύσουμε τα προβλήματα από τις Βρυξέλλες. Μπορούμε να στηρίσουμε τα εθνικά και περιφερειακά προγράμματα που αντιμετωπίζουν την κατάσταση, διότι διαφορετικά όταν υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι επενδύουν ε, στον ίδιο χώρο χάνεται το ενδιαφέρον βλέπω ότι εμείς έχουμε ε, κάτω από 2% ανεργία. Η στατιστική ότι έχουμε κάτω του 5% κάτω των 35 ετών δεν έχει σημασία διότι στο κοντινό μου χωριό ε, έχω νέους οι οποίοι μπορούν ε, να διαχειριστούν με τη νέα τεχνολογία εκμεταλλεύσεις 20 φορές μεγαλύτερες από ό,τι στο παρελθόν. Άρα πρέπει να δούμε την ποικιλομορφία της Ευρώπης και να αντιδράσουμε έτσι και όχι από τις Βρυξέλλες συλλήβδη με ένα κοινό μέτρο. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε να βρούμε λογικές ρυθμίσεις. Ευχαριστούμε Άλμπερτ, Άγνιου και μετά ο κύριος Κάπλος Αντός. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπερθεματίζω στα όσα είπε ο κύριο Ντες. Από τη μία μεριά λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει τον έλεγχο της παραγωγή και την άλλη λέει ότι χρειαζόμαστε νέους ανθρώπους στη γεωργία. Αυτά τα δύο δεν μπορούν να συμβαδίσουν. Και παρότι ο αριθμός των γεωργών επιχειρηματιών μειώνεται, η το εμβαδόν των ε, αγροτικών γεών στην Ευρώπη δεν μειώνεται. Το μόνο που έχει συμβεί είναι ότι σήμερα χρησιμοποιούμε γεωργικές μεθόδους που χρειάζονται λιγότερα εργατικά. Δεν χρειαζόμαστε τόσους ανθρώπους να εργάζονται στα αγροκτήματα όπως παλιότερα. Τα τρακτέρ γίνονται όλο και μεγαλύτερα και ούτω καθεξής. Ο λόγος για τον οποίο ασχολούνται μόνο μερικώς η ε, γεωργοί, απασχολούνται μόνο μερικώ. είναι ότι πριν από μερικά χρόνια είχαμε τα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία απαιτούσαν τέτοια εργασία, αλλά σήμερα όλα αυτά έχουν σταματήσει. Η καλλιεργία πατατών που γίνονταν ε, με τα χέρια, όλα αυτά έχουν σταματήσει πλέον. Κάτι Λείπει λοιπόν πιστεύω από την παρουσίαση όταν μιλάτε για το πώς μπαίνει κανείς, πώς ξεκινάει να γίνεται γεωργός. Ο καλύτερος τρόπος είναι να παντρευτεί μια εκμετάλλευση. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Αν είστε νέος και θέλετε, πολλά ζευγάρια έχουν κόρες και το έχω δει στη ζωή μου, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Και αυτό πιστεύω ότι έπρεπε να το συμπεριλάβει στην παρουσίαση, διότι συμβαίνει στην πραγματική ζωή. Υπάρχει κι άλλος ένας τρόπος για να μπει κανείς στη γεωργία, καθώς μεγαλώνουν σε ηλικία και δεν έχουν πλέον σωματικές κανότητες οι γεωργοί να κάνουν τις ε, εργασίες, ε, προσλαμβάνουν κάποιο νέο ο οποίος μαθαίνει σιγά σιγά τη δουλειά. Αυτό γίνεται στην Νέα Τώρα θα θέσω ένα δίλημα για τους τρεις ε, βουλευτές των Πρασίνων Πράγματι, από την αυξή της αγοράς εργασίας είχαμε μια ωφέλιμη κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον θάνατο δέντρων, διαφόρων δέντρων μέσω ασθενειών. Αυτά τα δέντρα πρέπει να ξαναφυτευτούν γρήγορα. Ωστόσο, θα πρέπει να ξαναφυτέψουμε δέντρα που δεν θα λαμβάνουν τις ίδιες ασθένειες, όπως οι βελανιδιές, οι λεύκες, γιατί να μην μεταφέρουμε. Να σας θυμίσω, πράσινοι φίλοι μου, δεν τρώμε δέντρα. Όσο λοιπόν ταχύτερα βάλουμε τα μυαλά μας να δουλέψουν για να έχουμε πιο ανθεκτικά δέντρα, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τους μυς μας για να τα φυτέψουμε. Αν θέλετε να επιχορηγήσετε ανθρώπους σε ε, περιοχές της βάλτε τους να κάνουν κάτι χρήσιμο. Ευχαριστώ. Bene, Agnew, adesso Luis. Ευχαριστούμε κύριε Άγνιο, κύριος Λουίς. Λουίς Καπλασάντος και μετά Σμιτ. Ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Ρεχίδορ για το έργο του και τη μελέτη του που είναι πολύ χρήσιμη σε αυτή τη φάση των διαπραγματεύσεων που βρισκόμαστε γιατί ήρθε η στιγμή να λάβουμε συγκεκριμένες ε, αποφάσεις ε, επί των προτάσεων που έχουμε ε, και συζητούμε. Και είναι πολύ χρήσιμο αυτό, ε, γιατί και στις γνωμοδοτήσεις μας ε, έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις ακριβώς για να δώσουμε ναύσματα σε νέους γεωργούς για να εισέλθουν στο επάγγελμα. Μην ξεχνάτε τις διαπραγματεύσεις που έχουμε στα πλαίσια του πρώτου πυλώνα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι βάσεις για μια συμβαστική λύση, ώστε το τόπα από των άμεσων ενισχύσεων που έχει προταθεί μόνο για τους νέους γεωργούς να επεκτείνεται και για τους νέους γεωργούς γενικώ, άσχετα με την ηλικία τους. Και αυτή την ερώτηση θέλω να υποβάλω στον καθηγητή Ρεχιδόρ. Δεν καταλήξαμε σε ένα ορισμό. Θα αφήσουμε στη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών να ορίσουν τον νέο γεωργό. Τον νέο εισερχόμενο δηλαδή. Γιατί ο νέο ερχόμενο γεωργό είναι κάποιο που για πρώτη φορά αναλαμβάνει γεωργική δραστηριότητα. Δηλαδή, δεν ήταν... αυτό σημαίνει ότι δεν ήταν ποτέ γεωργό ή πριν από 10 χρόνια είχε ασχοληθεί με τη γεωργία, μετά μεσολάβησε ένα κενό. Τα κράτη-μέλη θα βρουν τον ορισμό. Αλλά σίγουρα αυτό που μα ενδιαφέρει είναι να βρούμε ενάυσματα για του νέου γεωργού. Είτε είναι άνω είτε κάτω των 40 ετών. Είναι πολύ σημαντικό και χαίρομαι με τις προτάσεις ε, που τίνουν προ ένα συμβασμό προ αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, ω προ την πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, να βρούμε την σωστή ισορροπία μεταξύ μια κοινοτική πολιτική και μια εθνική πολιτική, όπω μα επισήμανε ο συνάδελφος Αλμπερντές. Δηλαδή δεν πρόκειται ουσιαστικά για μια εθνική πολιτική, αλλά μια ελαστικότητα που θέλουμε, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να εφαρμόσουν την πολιτική τους με βάση τις ιδιαιτερότητες εθνικές, στα πλαίσια όμως ενός κοινοτικού πλαισίου. Γιατί άλλες ε, ανάγκες έχουν ε, μερικέ περιοχέ και άλλες ανάγκες έχουν άλλε. Και σίγουρα στα πλαίσια της ανάπτυξη υπαίθρου δώσαμε αυτή την διακριτική ευχαίρεια και την ελαστικότητα στα κράτη-μέλη για να χρησιμοποιήσουν το α ή το β μέτρο. Βέβαια, ένα κράτος που δεν έχει πρόβλημα γύρασης των επιχειρηματιών του δεν χρειάζεται να αφιερώσει ιδιαίτερου πόρους στο μέτρο αυτό. Ένα άλλο κράτος όμως που έχει γυράσκοντα γεωργικό πληθυσμό σίγουρα θα δώσει προτεραιότητα στη χρήση αυτού του μέτρου. Ανάλογα με τις ανάγκες λοιπόν το, τα κράτη μπορούν να διαλέξουν τα εφαρμοστέα μέτρα. Ο κύριος καθηγητή καθηγητής έκρινε ότι οι προτάσεις είναι ανεπαρκείς σε ό,τι αφορά τους νέους επιχειρηματίες, όχι κατά ανάγκη γεωργούς. Όπως ξέρετε, η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπής που θα ε, στηρίξει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχεται τη δυνατότητα επενδύσεων και σε μη γεωργικέ δραστηριότητες. Ακριβώς για να προσελκύσουμε και άλλους οικονομικούς παράγοντες και άλλους ε, ε, εργαζόμενους που δεν είναι κατά ανάγκη γεωργοί. Απλώς θα εργάζονται στην Ήπεθρο. Νομίζω ότι αυτή είναι μια σωστή λύση πόλη δραστηριότητα, ώστε να εξασφαλίσουμε εισοδήματα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που δεν εξασφαλίζουν μόνο από τη γεωργία ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Είναι σημαντικό κάποιος γεωργός που ασχολείται με μερική απασχόληση να μπορεί να ασχοληθεί και με κάτι άλλο, να παραμείνει όμως στην Ήπεθρο και να εξασφαλίζει φυσικά ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Ευχαριστώ πολύ τον καθηγητή Ρεχιδόρ γιατί έδωσε απάντηση σε αρκετά ερωτήματα που μας ταλανίζουν. και ελπίζω ότι από τη μελέτη αυτή να βγουν αρκετές προτάσεις και στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις προτάσεις αυτές την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να δώσουμε λύση σε ένα πολύ σοβαρό και οξύ πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φάνηκε και από τα στοιχεία γιατί δείχνει πραγματικά μεγάλη γύρανση των γεωργών και ένα δάσος ε, χωρίς νέα δέντρα είναι ένα δάσος που είναι εξορισμού καταδικασμένο. Το ίδιο ισχύει μεταφορικά και για την γεωργία. Μία γεωργία που δεν θα ανανεώνεται με νέους γεωργούς δεν θα έχει μέλλον. Γι' αυτό και το συγκεκριμένη συνιστόση της κοινή γεωργικής πολιτικής θα έχει ιδιαίτερη σημασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Λουίς Σμιτ και μετά Ρούμπιξ. Κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαρίστως παρακολούθησα τον Λουίς ο οποίος μας εξήγησε πόσο ε, διεξάγονται οι συζητήσεις αλλά ήθελα να σας πω ότι την περασμένη εβδομάδα ήμουνα στην Βραζιλία και στην Παραγουάη και γι' αυτό με βλέπετε με τέτοια ενδυμασία σήμερα γιατί δεν έφτασαν τα πράγματά μου πίσω εν πάση περιπτώσει, έχουμε παρακολουθήσει τους ε, νέους γεωργούς και για μας το πρόβλημα είναι το ίδιο. Δηλαδή βλέπουμε με τι ενέργεια και ενθουσιασμό εκτελούν το επάγγελμά τους και κανείς ε, ε, δεν θα προσάψει κάτι στους νέους γεωργούς. Αλλά όταν μιλάμε για πρόσβαση και στη γη και την αποδοτικότητα η αγορά θα αυτορυθμιστεί και γι' αυτό πρέπει ε, ε, να κοιτάξουμε τις αιτίε και όχι για απλώς τα συμπτώματα διότι υπάρχουν προβλήματα σε ορισμένες χώρες και δεν νομίζω ότι θα πρέπει όλα αυτά να ρυθμιστούν σε γενικό επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ε, θέλω λοιπόν να ρωτήσω το φιλοξενούμενο μας. Οι, ιστορικές, τα ιστορικά δικαιώματα δημιουργούν και εκτιμένα και μήπως κάνουμε ε, λάθη ε, που βασίζονται στο, σε ιστορικές καταβολές και εμποδίζουμε νέους που θέλουν να μπουν στο επάγγελμα. Έχουμε πολλούς νέους στη Σκοτία οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν στη Γεωργία αργά. Μήπως έτσι αποκλείουμε την επόμενη γενιά των νέων γεωργών. Είναι ένα ουσιαστικό θέμα και δεν είναι ποτέ αργά να αλλάξουμε. Οπότε θα πρέπει να κοιτάξουμε πόσο πιο συχνά θα πρέπει να αναδιαμορφώνεται η δραστηριότητα, ποια θα είναι τα δικαιώματα, γιατί αυτό που με ανησυχεί είναι όποιος και να είναι ο συμβιβασμός και είμαστε στο σωστό δρόμο δεν θα αποδώσει διότι ε, δεν ασχολούμαστε με την αιτία παρά μόνο με τα συμπτώματα. Ενώ ο νέος πρέπει να δούμε αν μπορεί ε, να προχωρήσει και μπορεί να αποκτήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα αναγκαία. Δεν πρέπει δηλαδή να δεν θέλω να πω ότι ακολουθούμε κακή κατεύθυνση, αλλά δεν ε, ξέρουμε ακριβώς αυτά που θέλουμε. Ε, και κάποιος συμφώνησε με τον κύριο Άγνιο. ο κύριος Ρούμπιξ. Είμαι πολύ ικανοποιημένο Σας ευχαριστώ για αυτή την παρουσίαση. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Μα επέτρεψε να δούμε τι συμβαίνει στη Γεωργία σε ολοκλήρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ με τους συναδέλφους που μίλησαν πριν από μένα και ειδικότερα στο θέμα ότι δεν είναι δυνατό να διαχειριζόμαστε τα πάντα από τις Βρυξέλλες. Εγώ ίδιο εκπροσωπώ τη Λετωνία και συχνά Παρατηρώ ότι από εδώ στις Βρυξέλλες προσπαθούμε να ερθίσουμε πράγματα που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν καλύτερα σε εθνικό επίπεδο. Είπατε στην παρουσίασή σας ότι έχουμε τρεις επιλογές για την είσοδο στην αγορά. Κληρονομιά, δεύτερη επιλογή, ε, πρώιμη συνταξιοδότηση, εξαγορά δηλαδή από κάποιον άλλον και η είσοδος ως νέο εισερχόμενος εξ νόβο όπως είπατε εκ του μηδενός όπου πρέπει κάποιος να αναζητήσει γέες και δυνατότητες τώρα όσον αφορά την ανάληψη της εκμετάλλευσης ενός άλλου με την αλλαγή των γενεών ξέρω ότι στη Λετωνία έχουμε τη γεωργία ως παράδοση που μεταβιβάζεται στην επόμενη γενναία. Πάντα λοιπόν υπήρχε ένα κομμάτι του πληθυσμού που δούλευε στη γεωργία στο πλαίσιο οικογενειακών επιχειρήσεων. Στους σύγχρονους καιρούς σήμερα πλέον ε, δεν υπάρχει τέτοια συνέχεια, δεν υπάρχει τέτοια μεταβίβαση στην επόμενη γενναία. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν στη Λετωνία είναι ότι προσέζεται ένα πρόβλημα ε, ε, από αυτές τις πτυχές που σχετίζεται με τις κοινωνικές πτυχές επειδή οι πόλεις ε, σε αντίθεση με το αγροτικό περιβάλλον προσφέρουν πολλά περισσότερα στους νέους ε, ψυχαγωγία, υποδομές που υπάρχουν διαθέσιμες στις πόλεις και ούτω καθεξής. Η ερώτησή μου λοιπόν προς εσάς είναι έχετε μελετήσει το ποσοστό νέων αγροτών που κληρονομούν ε, γη, εκμετάλλευση από τους γονείς τους. Πώς είναι, σε ποσοστό. Ο κύριος και μετά κυρία Μαγκίνες. Στα πλέμα της πολιτικής ε, συνοχής ε, είδαμε και την πολιτική για τις πόλεις. εσείς καταλήγετε στο συμπέρασμα ότι στα πλαίσια της ΚΟΑ θα πρέπει να περιλάβουμε και την πολιτική της ε, υπαίθρου. Γιατί ασχοληθήκαμε με την πολιτική συνοχής ε, για την πολιτική στην ε, υπαίθρο. Αυτή τη στιγμή εντάσσεται στο δεύτερο πυλώνα. Θεωρείτε ότι είναι αρκετά τα μέτρα για την πολιτική της υπαίθρου γιατί πρόκειται για μια πολιτική που επηρεάζει το περιβάλλον και σχετίζεται φυσικά και με τις κλιματικές αλλαγές. Αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να είναι και αναπτυξιακή πολιτική η πολιτική της Υπέθρο, που, ε, μια πολιτική που θα υποστηρίζει την ε, ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων στην, στην Ήπεθρο, ενισχύοντας ε, την δυνατότητα των επενδύσεων. Οπότε μήπως θα πρέπει να προβλέψουμε κάποιες δραστηριότητες ε, στα πλαίσια και των εθνικών πολιτικών για να τονώσουμε την πολιτική της υπαίθρου, την πολιτική υπέρ της υπαίθρου. Στα πλαίσια της γεωργικής πολιτικής, ε, στα πλαίσια της πολιτικής ε, για τα τρόφιμα θα πρέπει έχουμε κοινέ εθνικές πολιτικές για τα θέματα αυτά. Γιατί να μην έχουμε κάτι αντίστοιχο και για την πολιτική της υπαίθρου. Να έχουμε και τέτοιες κοινέ πολιτικές για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Πιστεύετε λοιπόν ότι για την ανάπτυξη υπαίθρου θα είναι πιο πρόσφορες εθνικές πολιτικές εθνικέ πολιτικέ η μηπω θεωρειτε οτι θα πρεπει η δραση να αναλυθεί περισσότερο σε κοινοτικό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ε, ανάπτυξη τη υπαίθρου. Υπάρχει διαφορετική γεωργική ανάπτυξη στα κράτη-μέλη. Σε μερικές χώρες υπάρχει ένα πολύ ανεπτυγμένο σύστημα αγρομίσθωσης ε, που μάλιστα βρίσκει σύμφωνο και τους γεωργούς. Είναι πολύ ικανοποιημένοι από το σύστημα. Στη δική μου πατρίδα, για παράδειγμα, στην Πολωνία δεν έχουμε γενικευμένο σύστημα αγρομίσθωσης, ούτε ένα αρκετά τυποποιημένο σύστημα αγρομίσθωσης όπως σε άλλες χώρες. Οπότε, ανακύπτει το ερώτημα. Τι μέλη γενέστε, τι μπορούμε να κάνουμε για να μεταρρυθμίσουμε τη γεωργία και να αναπτύξουμε περισσότερο την ύπεθρο. Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ που εξετάζω αυτή τη στιγμή, θέμα που απασχολεί τους ε, συντάκτες της ε, γνωμοδότησης και για τις, οποίους, ε, και για τις οποίες καταθέτουμε πολλές τροπολογίες, πού πιστεύω ότι θα πρέπει να μας οδηγήσει, πώς θα μπορούσαμε να διορθώσουμε την κατάσταση στην, ε, και να βελτιώσουμε την ισχύουσα κοινή πολιτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω κάποιους νέους ε, γεωργούς που έχουν έρθει εδώ στη συνάντησή μας από την Ιρλανδία και τους καλωσορίζουμε και χαιρόμαστε που ακούν αυτή τη συζήτηση. Ήθελα απλά να πω ότι ο εισηγητής μόλις μίλησε για το έργο μας όσον αφορά τις τροπολογίες για τους νέους ε, γεωργούς και πιστεύω ότι πρέπει να στείλουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα μήνυμα υποστήριξης προς τους νέους ερχόμενους γεωργούς οι νέοι και οι εισερχόμενοι είναι δύο διαφορετικά είδη ε, γεωργών. Πρέπει να φροντίσουμε να λάβουμε μέτρα ώστε να βοηθήσουμε και τους δύο. Εδώ πρέπει να καταλαβούμε ότι μιλάμε για ανακύκλωση χρημάτων στη Γεωργία. Δεν υπάρχουν νέα χρήματα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτό το γεγονός. Κάποιες λοιπόν από τις πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες που παρουσιάζονται πρέπει να εξεταστούν υπό το πρίσμα των δημοσιονομικών περιορισμών που αντιμετωπίζουμε. Το επόμενο που θα ήθελα να πω σχετίζεται με το ζήτημα των διαφόρων προβλημάτων στα διάφορα κράτη-μέλη και ο συνάδελφος μου κ. Δες μίλησε για τη Βαβαρία όπου δεν υπάρχουν πραγματικά προβλήματα αλλά πρέπει να δούμε τι συμβαίνει πραγματικά και κάποια στιγμή πρέπει να δούμε τα κράτη-μέλη τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν δύο ενέργειες που οδηγούν σε αύξηση των τιμών των γεών και που θέτουν κάποια ζητήματα ανταγωνισμού στη Γεωργία και ίσως αυτή τη συζήτηση θα μπορούσαμε να την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Είναι παλιά τα νούμερα που παρουσιάζεται από το 2007 και εξακολουθούμε να έχουμε χαμηλό αριθμό νέων εισερχομένων αλλά στη χώρα μου ε, βλέπουμε την ε, αναγέννηση ενός νέου είδους γεωργίας. Πολλοί νέοι άνθρωποι μπαίνουν τώρα στον αγροδιατροφικό τομέα, ειδικότερα στο πλαίσιο της διατροφική ασφάλειας. Έχουμε κάτι νέο λοιπόν σε αυτό το τομέα που δεν διαφαίνεται στα νούμερα που αναφέρατε εσεί. Το τελευταίο που θα ήθελα να πω, τα σχόλια του κυρίου Άγγινς σε σχέση με το γάμο που πρέπει να κάνει κάποιο να παντρευτεί μια γυναίκα με αγρόκτημα αλλά ήθελα να πω ότι και οι γυναίκες ε, είναι γεωργοί και μάλιστα σε πολλά κράτη-μέλη λόγω των μικρότερων οικογενειών θα έχουμε όλο και περισσότερες γυναίκες οι οποίες θα κληρονομούν γη. είναι ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε πώς θα επηρεαστεί έτσι, η γεωργία και η παραγωγή τροφίμων. Η τελευταία παρατήρηση είναι βέβαια ότι στη χώρα μου ότι λένε ότι όπου υπάρχει θέλω υπάρχει και ένα συγγενής. Και συχνά όταν αποβιώνει ο ιδιοκτήτης ε, τρέχουν όλοι να κληρονομήσουν τη γη του. και υπάρχουν ευκαιρίες για όσους ενδιαφέρονται για τη Γεωργία να μπουν σε μια τέτοια επιχείρηση, σε τέτοιες περιπτώσεις. Και αν δεν υπάρχει επιχορήγηση για αυτούς είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεκινήσουν να ασχολούνται με αυτή τη δραστηριότητα. Και μία από τις ηχηρές απουσίες σε αυτή τη συζήτηση είναι ότι θα έπρεπε να έχουμε καλύτερες τιμές και υψηλότερα εισοδήματα ίσως να έχουμε ελάχιστα κίνητρα εισόδου ε, λόγω του χαμηλού επίπεδου των εισοδημάτων. Θα μπορούσαν να βελτιωθούν λοιπόν. Ευχαριστούμε Μαρία Τενάντζησία και μετά Καλινός. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή Ρεχιδόρ για την παρουσίαση της μελέτης που μας έκανε. Ήταν ε, πολύ χρήσιμη και ευχάριστη παρουσίαση. Ε, με προβλημάτισε πολύ αυτό που είπατε για την αντικατάσταση των ε, πιο ηλικιωμένων Γιώργων και δεν έχουν που να δώσουν τις κοιτάλοι. Μιλήσατε για τις ε, ζώνες 5Β. Ε, Εγώ είμαι από τη Ριόχα που ήταν ανέκαθεν ζώνα 5Β, γιατί ο στόχος των ζωνών 2 έφτασε πολύ αργά. Και μάλιστα εκεί ο συνδυασμός των τριών ταμείων λειτουργήσε πολύ καλά. Βέβαια, δημιούργησε πρόβλημα στους τεχνοκράτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον έλεγχο των ε, κονδυλίων. Γιατί αλλιώς δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί ήταν η πρώτη ζώνη που εξαφανίστηκε από την παλιά ταξινόμηση. Συμφωνώ ότι ο συνδυασμός των ταμείων με βάση τον h 5 ήταν πολύ χρήσιμος και λειτουργούσε και πολύ καλά. Άκουσα πολλούς νέους ε, Ισπανούς γεωργούς ε, να παραπονιόνται για ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ε, γιατί ιδιαίτερα για τους γεωργούς, περισσότερο από ό,τι για τους κτηνοτρόφους, ε, οι παλιοί γεωργοί πολύ απρόθυμα εγκαταλείπουν δραστηριότητα γιατί έχουν πάντα το δέλεαρ των κοινοτικών ενισχύσεων. Αυτοί που εγκαταλείπουν τη γεωργική δραστηριότητα θα πρέπει να σταματούν φυσικά να λαμβάνουν τα, τα, τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής ε, Γεωργικής Πολιτικής και αυτή την προσπάθεια κάνει ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαχωρίσει σαφώς τους ενεργούς γεωργούς από του ε, μη ενεργού, ε, Θέλουμε να ορίσουμε τι εστί ενεργό γεωργός και να καταλήξουμε σε ένα δόκιμο ορισμό ώστε να μην αποκλείσουμε κανέναν ενεργό γεωργό αλλά να μην ωφελήσουμε κανέναν που κρατά μόνο τους τίτλους της γη για να εξακολουθεί να έχει πρόσβαση στα κονδύλια παρόλο που έχει καταλήψει τη γεωργική δραστηριότητα. Αυτό είναι άδικο για του νέου ειδικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε για τους απασχολούμενους στην Ήπεθρο γενικώ, άσχετα με τη γεωργία. Το θέμα τη πολυλειτουργικότητα ήταν πολύ σημαντικό. Παλιότερα δεν είχαμε αρκετά χρήματα για άμεση ενισχύσει προ του γεωργού και του κτηνοτρόφου και τότε εφεύρε την ωραία λέξη πολυλειτουργικότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πει ότι όσοι ασχολούνται και με άλλε δραστηριότητε πριν τη γεωργία και τη κτηνοτροφία ε, θα μπορούσαν ε, να συμπληρώσουν το εισόδημά του για να συνεχίσουν τι γεωργικέ δραστηριότητε. Και με αυτή την πολυλειτουργικότητα μερικοί συμπλήρωσαν το γεωργικό της εισόδημα με τουριστικές δραστηριότητες ή με άλλες δραστηριότητες αναψυχής. Αν δεν προσέξουμε στον ορισμό του ενεργού γεωργού, ίσως βλάψουμε τους γεωργούς. Γιατί αυτό ήταν το κληροδότημα της προηγούμενης μεταρρύθμισης ΚΑΠ. Ε, που πρόθεσε με ιδιαίτερο μένος η κυρία Φίσερ Μπόλ, προηγούμενη επίτροπος. Προσοχή λοιπόν να μην αδικήσουμε τους Γιώργους, προσοχή σε αυτόν τον ορισμό. Σε ό,τι αφορά τη βοήθεια της επιδοτής που προτείνεται στους απασχολούμενους στην Ήπειθρο Γενικό, αυτό με φοβίζει κάποιος, γιατί έχουμε πολλούς που απασχολούνται στην Ήπεθρο και δεν ασχολούνται με γεωργικές δραστηριότητες. Και μάλιστα σε μερικές χώρες που είναι πολύ ανεπτυγμένε οι τεχνολογίε πληροφορική. Υπάρχουν άνθρωποι που διαμένουν στην Ήπεθρο και ασχολούνται με την πληροφορία και δεν έχουν λοιπόν καμία σχέση με τον πρωτογενή τομέα. Προσοχή λοιπόν, μην αφιερώσουμε ενισχύσεις της ΚΑΠ σε απασχολούμενο στην Ήπεθρο που δεν έχουν καμία σχέση όμως ούτε με τη γεωργία, ούτε με την κτηνοτροφία, ούτε γενικώ με τα χωράφια. Απλώς ασχολούνται με άλλες δραστηριότητες και διαμένουν στην Ήπεθρο και θα αντιμετωπίσουμε και πρόβλημα νομικής βάσης γιατί οι επιδοτήσεις αυτές ε, έχουν συγκεκριμένο σκοπό να στηρίξουν τον πρωτογενή κλάδο. Προσοχή λοιπόν αν ε, διοχετευτούν σε άλλες δραστηριότητες. Άλλωστε για άλλους τομείς οι επιχειρηματίες ε, δικαιούνται επιδοτήσεις από άλλα κεφάλαια του κοινωτικού προϋπολογισμού. Δεν είναι ανάγκη να τα πάρουν από τη Γεωργία. Ο κύριος Καλινόφσκι και τελευταίος ο κύριος Δαντά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή για την ανάλυση που μας έκανε και να αναφερθώ σε τρία θέματα. Το πρώτο αφορά ένα θέμα που πολύ ακροθυγώς ε, το θίξατε κύριε, ε, προ, κύριε καθηγητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 7% των γεωρικών ε, γεών για οικολογικούς σκοπούς. Ε, αν όμως ε, όντως υιοθετηθεί αυτό το ποσοστό, θα πρέπει να αυξηθούν οι εισαγωγές των γεωρικών προϊόντων. Ιδιαίτερα σε κάποιες μικρές περιοχές που εξορισμού είναι οικολογικού ενδιαφέροντος τόπερ. Οπότε θα χρειαστούν ε, εισαγωγές των γεωρικών προϊόντων. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας προτείνει μείωση της ε, παραγωγής βιοκαυσίμων πρώτη γενιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ ασυνεπής αυτή η πρόταση και δεν θα έχει κανένα θετικό αποτέλεσμα. Δεύτερο θέμα, το πρόγραμμα, το καθεστώς για του μικροκαλλιεργητέ. Εγώ είμαι Πολωνός. Εκεί έχουμε ε, πραγματικά κατακαιρματισμό των γεωργικών γεών και τέτοιο καθεστώς ε, για τους μικροκαλλιεργητές θα είναι ωφέλιμο κυρίως για τις χώρες που έχουν ε, πολλούς μικροκαλλιεργητές και μεγάλο κατακαιρματισμό των γεωργικών εκτάσεων. Και πιστεύω ότι θα είναι πολύ θετικό αυτό το πρόγραμμα και το καθεστώς, αλλά δυστυχώς με τη μορφή του έχει, πολύ φοβάμαι ότι θα έχει περισσότερα αρνητικά παρά, θετικά αποτελέσματα. Και θα σας δώσω ε, ένα ε, παράδειγμα. Έχουμε σήμερα το 20%, 7 εκτάρια, για τους, ε, για, 7 εκτάρια και κάτω για τους πολωνικούς όρους, περίπου δηλαδή 70% του συνόλου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Πολωνία εμπίπτουν στον, στον, στην κατηγορία αυτή. Βέβαια, ε, οι, μισοί, οι μισές τέτοιες εκμεταλλεύσεις δεν ε, έχουν πραγματικά γεωργικό προσανατολισμό. Και αν ε, ενταχθούν σε αυτό το, στο πρόγραμμα θα λαμβάνουν γεωργικές ενισχύσεις χωρίς να έχουν καμία γεωργική δραστηριότητα. Επιπλέον το σύστημα αυτό προτείνεται ώστε κάποιος άσχετα αν έχει ένα, πέντε ή εφτά εκτάρια να λαμβάνει ένα καταποκοπή ποσό. Ένα καταποκοπή ποσό ισχύει για όλους, άσχετα με το εμβαδόν της γεωρικής εκμετάλλευσης. Οπότε, αυτό που σήμερα έχει ένα εκτάριο και παίρνει σήμερα 20 ευρώ και αυτό που έχει 7 εκτάρια και σήμερα στην Πολωνία λαμβάνει 1.400 ε, ευρώ, με το νέο σύστημα θα πάρουν και οι δύο και ο πρώτος και ο δεύτερος 800 ευρώ. Δηλαδή γίνεται μια εξημείωση άσχετα με το εμβαδόν της ε, γεωργικής έκτασης. Αυτό πραγματικά είναι άρρωστο, είναι άδικο. Οπότε Ποια είναι η νομιμοποίηση αυτής της μεταρρύθμισης. Θα έχει τα αντίθετα από τα ανανεώμενα αποτελέσματα. Και πώς θα ξέρουμε ότι οι γεωργοί δεν θα κατακαιρματίσουν εσκεμμένα τις εκμεταλλεύσεις ώστε να λαμβάνουν περισσότερες ενισχύσεις. Από τη στιγμή που η ίδια ενίσχυση κατά ποσό θα ισχύει είτε για ένα, είτε για δύο, είτε για 7 εκτάρια. Και τι, υπάρχουν και γεωργοί που δεν καλλιεργούν τη γη, καλλιεργούν μόνο τον, τρόπο απορρόφησης κονδυλίων. Είναι απαράδεκτο να ενισχύουμε ε, ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με τη γεωργία, που δεν ασκούν καμία γεωργική δραστηριότητα. Επίσης, μιλήσαμε για την επιδότηση νέας επιχείρησης ε, στη γεωργία, το startup. Στην ε, Πολωνία έχουμε ενιαία πληρωμή άσχετα με την ε, με το εμβαδόν της γεωργικής έκτασης. Τώρα, αν έχουμε ένα, ένα νέο σύστημα, ένας νέος που θέλει να αρχίσει η δραστηριότητα, μπορεί να θέλει να επεκτείνει ε, την ε, επιχείρησή του προς τον γείτονα, που δεν έχει γεωρική δραστηριότητα, αλλά έχει δικαίωμα να λαμβάνει ενισχύσεις. Οπότε ε, θα μπορέσει να αγοράσει το τη γειτονική εκμετάλλευση, αλλά εδώ δεν υπάρχει διάκριση και δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ο Γιώργος που λαμβάνει την εκμετάλλευση όντω ασκεί γεωργική δραστηριότητα. Μήπως λοιπόν μπούμε με τα νέα μέτρα σε ένα τούνελ που όχι μόνο θα αποτρέψουμε τους ε, γεωργούς, τους νέους γεωργούς να ασχοληθούν με τη γεωργία, αλλά θα έχουμε όλο και περισσότερη γεωργική παραγωγή και θα απειληθεί και ο ίδιος ο ανεφοδιασμός μας σε τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή. Ωραία, ευχαριστούμε κύριε Καλινόφσκι, κλείνει ο Ντάντα και μετά ο κύριος καθηγητής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά για την παρουσίαση. Έχω δύο ερωτήσεις και ένα σχόλιο. Οι ερωτήσεις πρώτα. Στις προπαρασκευαστικές εργασίες που διεξάγατε, ασχοληθήκατε με κάποια ανάλυση αναχώρα όσον αφορά τα εργαλεία τα οποία υλοποιήθηκαν και συγκρίνατε την αποτελεσματικότητα αυτών των εργαλείων. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη μου ερώτηση σχετίζεται με τα όσα ανέφεραν ο κ. Αλμπερντές και ο Ζεζεμποβέ όσον αφορά τι περιφερειακές ιδιαιτερότητες και το γεγονό ότι σήμερα μια επαγγελματική γεωργική εκμετάλλευση στι περισσότερε χώρε μα απαιτεί σημαντικά κεφάλαια. Έτσι λοιπόν, ένα από τα προβλήματα τη γεωργία είναι η πολύ χαμηλή απόδοση των κεφαλαίων και η ανάγκη τελικά μακροπρόθεσμη επένδυση. Δεδομένη αυτή τη κατάσταση που διαρκώ αμβλύνεται διότι είναι όλο και μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις σε όλες τις χώρες ε, στη... κατά την εργασία σας μήπως ε, βρήκατε κάποιες ιδέες που θα μπορούσαν πέραν των όσων μας προτείνατε σήμερα να απαντήσουν σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα του κεφαλαίου που είναι απαραίτητο για την εκμετάλλευση. Και τελευταίο ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, νομίζω ότι υπογραμμίσατε στην εισαγωγή, ανεξαρτήτως των καταστάσεων στις τοπικές κοινωνίες που γνωρίζουμε όλοι. Εάν ε, μόνο 6% είναι οι κάτω των 35% γεωργοί ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 4,5 εκατομμύρια είναι άνω των 60 ετών. Παρότι δεν είναι ακόμα ορατό, υπάρχει περίπτωση ερήμωσης στο μέλλον πολύ μεγάλων περιοχών εάν δεν φροντίσουμε να αντικαταστήσουμε αυτούς τους γεωργούς τα εργαλεία της ΚΑΠ σήμερα επιτρέπουν σε όλες τις χώρες να κάνουν κάτι ελάχιστες όμως χώρες έχουν υλοποιήσει συγκεκριμένες πολιτικές ε, για την εγκαθιδρύση των εισερχομένων Ωραία, ευχαριστούμε όλους ε, για τα σχολιά τους. Ξαναδίνω τώρα το λόγο στον ε, καθηγητή κύριο Χεσούς Κονζάλης ε, για να απαντήσει, αλλά δυστυχώς κύριε καθηγητά πρέπει να απαντήσετε σε 10 λεπτά γιατί διαφορετικά θα μας εγκαταλείψουν οι διερμηνείς μας. Ευχαριστώ. Δέκα λεπτά χρειάζομαι μόνο και μόνο για να συνοψίσω τις ερωτήσεις δεν μου δίνεται αρκετό χρόνο, θα πρέπει να αυτοσχεδιάσω λίγο την απάντηση. Πάντως υπάρχουν τρία-τέσσερα ζητήματα που καλό θα ήταν να τα επισημάνουμε. Το πρώτο το επισήμανε ο τελευταίος ομιλητής, ότι δεν υπάρχουν νέοι γιατί δεν φεύγουν οι παλιοί. Οι νέοι είναι το 15% μόνο της ιερικής απασχόλησης, ενώ οι πιο ηλικιωμένοι πάνω από 40% υπάρχει το στοιχείο στην έκθεση. Και έχουμε 20 και πίνακες με τα διεξοδικά στοιχεία χώρα. Θα τα λάβετε στην οριστική, έκθεση, στην οριστική μορφή της έκθεσης. Πολύ σημαντικό επίσης είναι και το θέμα ότι υπάρχουν οικονομικοί λόγοι, πολύ σημαντικοί οικονομικοί λόγοι, ώστε οι πιο ηλικιωμένοι να μην εγκαταλείπουν τη γεωργική δραστηριότητα. Υπάρχουν λόγοι για του οποίου παραμένουν στη γεωργία οι πιο ηλικιωμένοι γεωργοί. Γιατί ε, με τι ενισχύσει που λαμβάνουν του συμφέρει να παραμείνουν παρά να συνταξιοδοτηθούν. Γι' αυτό και δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν τη Γεωργία, γιατί μπορούν να συνεχίσουν ε, επαόριστο να λαμβάνουν τι κρατικές, τις ε, γεωργικές ενισχύσεις. Κάποιες χώρες, όπως η Γαλλία για παράδειγμα, ε, θα καταστήσουν ασύμβατες τις γεωργικές ενισχύσεις με τις συντάξεις. Δεν ξέρω αν το έχουν εφαρμόσει. Πάντως ε, αυτή η ασυμβατότητα δεν ε, χρησιμεύει αυτή τη στιγμή για να στείλει σε συνταξιοδότηση τους Γιώργους. Κάποιος βροβουλευτής από τη Γερμανία είπε ότι δεν θα πρέπει όλα να τα ρυθμίζουμε κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, θα συμφωνούσα αν είχαμε μια πραγματικά ισχυρή γεωρική πολιτική. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ε, αμφισβητείται ο πρώτος ε, πυλώνας, αλλά ο κύριος ε, από τη Γερμανία δεν μίλησε για τον πρώτο πυλώνα, μίλησε για την μειοψηφία, για το δεύτερο πυλώνα. Ο δεύτερος πυλώνας όμως, αν αφήσουμε τις αμυγείς πολιτικές, αγροεπιστηστικό τομέα δηλαδή και αγροπεριβαλλοντικό, ουσιαστικά μένει ένας πολύ μικρός πυλώνας. Μένει μια κολονά, ένα κολονάκι ουσιαστικά ο πυλώνας, ο δεύτερος. Αν αφαιρέσουμε τα αγροεπιστηστικά και τα αγροπεριβαλλοντικά, είναι 15% της συνολικής ΚΑΠ. Οπότε αυτό το τμήμα που είναι ύπεθρος και όχι γεωργικό, είναι το 10% του 15%. Μιλάμε για 1,5% ουσιαστικά. Οπότε δεν έχουμε μια ισχυρή πολιτική, αγροτική πολιτική, πολιτική της υπαίθρου στην Ευρώπη. Δεν βλέπω λοιπόν τον κίνδυνο που επισήμανε ο κύριος ο Ευρωβουλευτής από την Γερμανία. Η Γερμανία και άλλες χώρες έχουν πολύ ισχυρές δικές τους πολιτικές για την Ήπεθρο. Και η Γερμανία και η Γαλλία έχουν ισχυρές πολιτικές για την Ήπεθρο. Το ίδιο και οι κατοχώρες, οι σκανδιναβικές χώρες. Η Ισπανία το προσπάθησε αλλά δεν τα κατάφερε. Έχει τον νόμο <laughs> αλλά δεν έχει τα χρήματα. Οπότε τι συμβαίνει. Η αγροτική πολιτική, η εθνική πολιτική για την Ήπεθρο είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να ενισχυθεί όμως. Αλλά όχι ο καθένας όπως του κατέβει. Όχι ο καθένας όπως το σκεφτεί για να μην έχουμε αντίφαση μεταξύ των κρατικών, των κρατικών των εθνικών μέτρων και των κοινοτικών. Θα πρέπει να έχουμε ένα κοινοτικό πλαίσιο, όχι υπερβολικά σχολαστικά κοινά μέτρα, αλλά πόσα άρθρα έχει ο γαλλικός ιερικός κώδικας, 300 και. Θα μου πείτε ότι είναι περίπλοκη η πολιτική. Στην τελευταία μεταρρύθμιση, αν δεν κάνω λάθος, αναθεωρήθηκαν 125 άρθρα πολύ περισσότερο δηλαδή από ότι ο κανονισμός για την ανάπτυξη πέθρου. Οπότε τι λέμε εδώ. Χρειαζόμαστε μία συνέπεια, μία συνοχή μεταξύ των διαφόρων διατάξεων. Επίσης ε, είπαμε να δούμε αν μπορέσουμε να ενισχύσουμε τη... τους νέους ερχόμενους. Αντιλαμβάνομαι τα ε, σχόλια και τα χαριτολογήματα του Βρετανού συναδέλφου. Το βλέπουμε μερικές φορέ και στι ταινίε, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Στην ε, Ισπανία και στην ε, Μεγάλη Βρετανία έχουμε ελάχιστο ποσοστό ε, εξαγοράση συνέχιση. Στη Γερμανία έχουμε μεγάλο ποσοστό, 100. Ενώ άλλε χώρε, οι χώρες της Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, σε χαμηλό ποσοστό. Το ίδιο και το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν υπάρχει διαδοχή, δεν υπάρχει αντικατάσταση. Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν δεν έχουν ε, σε που να δώσουν τη σκητάλη μερικοί γεωργοί. Επίσης, ε, δεν είναι ότι έχουμε μια τομεακή προσέγγιση του προβλήματος. Γιατί όσοι ασχολούμαστε με τη γεωργική οικονομία, με την οικονομία της υπαίθρου, έχουμε συνηθίσει σε φράσεις ε, «δεν υπάρχει τίποτα χωρίς γεωργία», «δεν γίνεται τίποτα χωρίς τη γεωργία». Είναι αλήθεια μεν, αλλά όλο και λιγότερο αλήθεια γίνεται μια τέτοια διαπίστωση. Η γεωργία είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, δεν το αφισβητεί κανεί, αλλά σε πολλέ ε, περιοχέ και ζώνε ε, και άλλε δραστηριότητε που δεν είναι απλώ συμπλήρωμα τη γεωργία, είναι πραγματικά ξεχωριστέ αυτοτελεί δραστηριότητε που επίση είναι απαραίτητε για την επιβίωση τη γεωργία. Και είναι πολύ σημαντικό να στηρίξουμε και αυτέ τι δραστηριότητε. Οπότε λέτε και από πού θα προέλθουν όλα αυτά. Ο φόβος της Ισπανίδας συναδέλφου. Από πού θα χρηματοδοτηθούν όλα αυτά. Γνωρίζω ότι κάθε φορά που κάποιος φοβο τη ισπανιδα συναδελφου απο διάλεξη, κάποιος καποιο δινει διαλεξη καποιο απο τα συνδικάτα σηκώνει το χέρι και λέει όχι αφήστε κάτω τα χρήματά μας. Τα συνδικάτα θεωρούν ότι είναι οι μοναδικοί δικαιούχοι των κονδυλίων της ΚΑΠ. Αλλά αυτό δεν είναι απάντηση. Γιατί θα μπορούμε να πούμε στα γεωργικά συνδικάτα και εσείς τι κάνετε με την ανάπτυξη πέθρου. Γιατί και αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Αν δεν μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε την ύπεθρο με την ΚΑΠ, θα πρέπει να βρούμε άλλα κονδύλια ή με εθνικά κονδύλια και επίσης κοινοτικά. Το θέμα είναι ότι αν χρειαζόμαστε ένα κοινοτικό πλαίσιο, χρειαζόμαστε και κοινή χρηματοδότηση, κοινοτική χρηματοδότηση. Υπάρχουν κονδύλια, αλλά είναι εγκατασπαρμένα, είναι στο Φεντέρ, ε, σε μία ζώνη ε, διορθώνεται η γέφυρα, αλλά δεν διορθώνεται ο δρόμος. Οπότε έχουμε ουσιαστικά μία, ένα κατακαιρματισμό των κονδυλίων και μία ε, διάχυση που δεν έχει αποτελέσματα, γιατί δεν υπάρχει συγκέντρωση και τελικά κάνω μια τρύπα μέσα στο νερό. Και γι' αυτό θέλουμε να διορθώσουμε την κατάσταση το και να επανέλθουμε στο 2020 σε ένα μέτρο που εφαρμόζαμε το 1999. Βλέπετε με τι ρυθμούς ε, εκτελούμε τις μεταρρυθμίσεις. Και τέλος, προσοχή με τις ε, βοήθειες προς τις μικρές και τις μεγάλες καλλιέργειες, τις μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Θα διαπιστώσετε από τους πίνακες ότι ε, στις χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ε, το μέσο, ο μέσος όρος των κρατικών ενισχύσεων είναι πάνω από 200.000 ευρώ. Ενώ για τις παλιές χώρες το 2015 είναι πολύ χαμηλότερα τα ποσοστά. Στη Γαλλία, στη Γερμανία, ένας εμπειρογνώμας μου είπε όμως μην ε, μπερδεύεσαι γιατί είναι συνεταιρισμοί. Όλοι είναι συνεταιρισμοί, δηλαδή όλοι είναι γεωργικοί συνεταιρισμοί για να φτάσουν στο 200.000 κατά μέσο όρο ευρώ αναδικαιούχο ή μήπως έχουμε μια ραγδαία συγκέντρωση των ενισχύσεων, των γεωρικών ενισχύσεων σε λίγα χέρια στις χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπως είχαμε αρχικά το φαινόμενο στις προηγούμενες παλιές χώρες. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια τεράστια συγκέντρωση των γεωργικών ενισχύσεων και φάνηκε αυτό και από ένα πίνακα. Είναι γνωστά όλα αυτά. Και όταν λέμε ότι θα βοηθήσουμε τις μικρές και τις μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τι, τι να κάνουν, τι να κάνει κανείς με 500 ευρώ. Δεν μπορεί να ζήσει κανείς με 500 ευρώ. Ευτυχώς ε, έχει και άλλα έσοδα. Αλλά δεν θέλουμε να εγκαταλείψει τη γεωργία. Γιατί πολλά, σε πολλά εδάφη αυτή η μικρή εμβέλεια γεωργίας μαζί με άλλες δραστηριότητες υπαίθρου είναι απαραίτητες και για την τοπική οικονομία αλλά και για το περιβάλλον και για την ε, περιοχή ευρύτερα. Οπότε έχουμε διάφορα στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Λυπούμε που μακρηγορώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω να διευρύνετε λίγο τους ορίζοντες. Yeah. Ίσως θα πρέπει μια πολιτική της υπαίθρου να τη μοιράσουμε. Ένα τμήμα να εμπίπτει στην ΚΑΠ και άλλο τμήμα να εμπίπτει σε άλλες πολιτικές που θα πρέπει να τις ε- επαναφέρουμε στην Ήπεθρο. Να έχουμε μία, ε, μία άμυλα μεταξύ ε, της, των πόλεων και της πολιτικής για τις πόλεις και της, της πολιτικής για την Ήπεθρο. Γιατί Παλιά δεν είχαμε την ε, ύπεθρο μόνο στην ΚΑΠ. Στο παρελθόν είχαμε ένα πολύ σημαντικότερο τμήμα της υπαίθρου στη συνοχή. Με τις μεταρρυθμίσεις ξεφύγαμε από τη συνοχή και περιορίσαμε την ύπεθρο μόνο στην κοινή γεωρική πολιτική. Και προβληματιζόμαστε τώρα με την αλλαγή γιατί ακριβώ ε, συζητούμε τη μεταρρύθμιση. θα πρέπει να περιμένουμε άλλη μια αίτια για να το ξαναθέσουμε και μερικοί δεν θα είμαστε καν ζωή, ή δεν θα είμαστε καν στο επάγγελμα για να μπορούμε να επισημαίνουμε όλα αυτά τα θέματα. γράφια, σε ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσία σα Όλα αυτά είναι επιχειρήματα και θέματα που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει η Κομισιόν μα, η Επιτροπή μα με όλο και στενότερα περιθώρια μάλιστα. Είναι πιεστικά τα περιθώρια. Έτσι θα επιταχύνουμε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ όσους ε, μίλησαν. Υπενθυμίζω αύριο στι 9 η ώρα για... θα συναντηθούμε στο Συμβούλιο στι 9 η ώρα με του ηγητέ και του κοιόδη. Η Επιτροπή καλείται για τι 10 και 4. Ελπίζουμε ότι 10 και 4 θα έχουμε ολοκληρώσει το πρώτο κομμάτι. Ευχαριστώ όλους και καλό βράδυ.